Merci, madame. Πρόεδρε Σαρτουή, σα ευχαριστώ κύριε μου. Και τώρα θα υποβληθούν οι ερωτήσει με την εξή μέθοδο. Δύο διαφορετικέ μέθοδοι. Πρώτα-πρώτα θα τοποθετηθούν οι πολιτικέ ομάδε. Η κάθε μία θα τοποθετηθεί με κάποιον αγορητή και κατόπιν σε μία δεύτερη ερωτήσεων θα τεθούν ερωτήσει πρώτα-πρώτα σε σχέση με τον προπολογισμό, στη συνέχεια δε με τον έλεγχο του προπολογισμού. Τέλο δε ερωτήσει σε σχέση με ε, νομικά ζητήματα. Ο πρώτο ο οποίο θα λάβει το λόγο όσον αφορά την πρώτη σειρά ερωτήσεων θα είναι ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να συγχαρώ την ε, υποψηφία Επίτροπο. Έδειξε τις ικανότητές της, έδειξε την πείρα της με αυτή την εισήγηση. Έδειξε επίσης ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα του προπολογισμού και γνωρίζει και αυτά τα οποία μας απασχολούν. Αναφέρατε κυρία, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τι πληρωμέ. Πετε μα εσεί, τι προτίθεστε να κάνετε εσεί, τι δέσμευση να λαμβάνετε σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Πώ θεωρείτε ότι θα σταθεροποιήσετε την κατάσταση, πώ θεωρείτε ότι θα επιλύσετε το πρόβλημα. Υπενθυμίζω ότι το 2014 είχαμε κρεμούσε πληρωμέ ανά των 23 δι και τέλη το έτο θα έχουμε δεκάδε ε, επίσης χιλιάδων ε, ευρώ τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν και παραπάνω. Εσείς ε, τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε τόσο ώστε να μην απολέσουμε την αξιοπιστία την οποία τόσο χρειαζόμαστε. Γεωργίευα. Σας ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και πάρα πολύ επίκαιρη. Είναι κάτι το οποίο όλους μας απασχολεί. σε τρεις άξονες θα μπορούσαμε να απαντήσουμε. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ε, εξυπηρετήσουμε τις οφειλές που ήδη έχουμε σωρεύσει. Δηλαδή, αλλιώς θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την, το σχέδιο που προϋπορίζουν το 2014 και την ευελιξία που θέλουμε να επιφέρουμε όσον αφορά το αποθεματικό για τα κατεπίγοντα Και αυτές είναι προτάσεις που ισχύουν για αυτή τη χρήση και για την επομένη του χρόνου. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και επίσης ε, ελπίζω να μπορέσουμε να την βελτιώσουμε. Βέβαια. Δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα αρκεστούμε σε αυτά. Και εδώ έρχομαι τώρα στο δεύτερο άξονα της μεθόδου μας ε, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σωστή διαχείριση, τι θα κάνουμε προγράμματα και έργα, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτά να τα εκτελέσουμε ε, με επιτυχία. Όπως ξέρετε, ήδη το ξεκινήσαμε αυτό σε όλους τους τομείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ίδια το, το έκανα αυτό και το και ένιωσα την ανάγκη να γίνει αυτό στην ανθρωπιστική βοήθεια. Εκεί έπρεπε να πετύχουμε οπωσδήποτε και να μην έχουμε κανένα είδου ε, συγκρούσει, αντιφάσει, ε, αποτυχία. Τέλο πάντων, η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να ατενίζουμε το μέλλον. Το έχουμε υπόψη τι θα κάνουμε και αν λέμε ότι με τι δεδομένε προκλήσει τι θα κάνουμε, πώ θα ε, προσεγγίσουμε ε, το, τα θέματα του κοινωτικού προπολογισμού, ε, να προβλέψουμε την κατάρριξη των προσπαθειών μας, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνουμε αυτό το οποίο εσείς είπατε, δηλαδή, δηλαδή πρόθεσμα να ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτών των δυσκολιών που έχουμε σε σχέση με τις πιστώσεις των πληρωμών. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριο, η κυρία, συγγνώμη, Γκάρντια Θάβαλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Υπόψηφη Επίτροπε, κυρία Γεωργίευα μας μιλήσατε στην εισήγησή σας όσον αφορά ε, το δημοσιοκοπλαίσιο, πλαίσιο, μιλήσατε και για αυτήν την mid-term review, ε, αυτή τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λόγια εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και εμεί θέλουμε να κάνουμε μια μετεκλογική αναθεώρηση. Γι' αυτό πρόκειται τώρα να μα καίει κατά αυτή τη θητεία. Οπότε θα θέλω να μου πείτε εσεί τι θα κάνετε θα ξεκινήσετε αυτή την μετεκλογική αναθεώρηση, θα λάβετε υπόψη την πρόταση Γιούγκερ σε σχέση με το πρόγραμμα επενδύσεων των 300 δις. Ε, θα λάβετε μέρος σε αυτή την ομάδα συντονισμού αυτού του σχεδίου, του προγράμματος επενδύσεων. Ε, τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά τα 300 δις στον κοινωτικό προϋπολογισμό. Είναι πρόκειται για την πρόταση Γιούγκερ. Εσείς, εσείς καθώς σας αναλογεί τι διαχείριση θα κάνετε, επίσης τι μέσα, τι εργαλεία θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχετε, ούτως ώστε να μπορέσετε να πετύχετε στο έργο σας. Γεωργίου. Σας ευχαριστώ. Δύο σκέλη ερώτησή σας, να απαντήσω ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα. Ως μέλος αυτής της Επιτροπής είμαι υπέρ του να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε και τις δεσμεύσεις, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κατά τις διαπραγματεύσεις, προς το Κοινοβούλιο δεσμευθήκαμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό τον επταετή προγραμματισμό και να μην ξανασχοληθούμε μαζί του. Και πρόκειται για έναν κόσμο που αλλάζει άρδεν. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί κανείς να προβλέψει με έναν ορίζοντα επταετίας τι θα γίνει με κάποιον προϋπολογισμό που τώρα καταρτίζεται διότι συνεχώς έχουμε αλλαγές και αλλαγές σημαίνουν ότι θα πρέπει κανείς να μπορεί μέσω πρόθεσμα να κάτσει να αναθεωρήσει να δει ε, τι γίνεται με το πολιετές πλαίσιο σε την κατάσταση, τη συγκυρία θα από τις οικονομίες μας, πώς θα τα πηγαίνουμε, πόσο εκτελούμε τους, τους προϋπολογισμούς, ποιες είναι οι, οι προτεραιότητες ανά πάσα στιγμή και να δούμε πώς θα τα πάμε. Όμως είμαι αφοσιωμένη σε αυτό τον στόχο και παίρνω πολύ σοβαρά το ρόλο μου τώρα για το δεύτερο σχέδιο της ερωτήσεως. Τι λένε, είπατε. Ότι εξετάζεται ξετινάζετε τους υποψηφίους επιτρόπους και ίσως ο συνάδελφος ο Αρμόδιος θα σας πει για αυτά τα 300 δις στο πακέτο αυτών των επενδύσεων. Και βεβαίως έχουμε τις παραμέτρους της συνεργασίας και ο δικός μου ρόλος είναι το να μπορέσουμε με τον προϋπολογισμό να δημιουργήσουμε, να ελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις. Σας είπα για τη μόχλευση τριπλασιάσαμε τα σχετικά με τα χρηματοδοτικά όργανα και εργαλεία. Και υπάρχει για τις ε, ΜΜΕ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ αξιόλογο και θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει κεφάλαιο για αυτές, μια πρικοδότηση για να μπορέσουν να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι και η μόχλευση αφορά μια αναλογία 1 προς 5. Και αυτό έχει σχέση άμεσα με τις επενδύσεις, οπότε θα πρέπει να κάτσουμε και να τα ζυγίσουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά ή να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. αυτό είναι ε, η προτεραιότητά μου. Εμένα, αλλά και των άλλων επιτρόπων και συμπαθάτε με που επερεύει τον χρόνο. Θα πρέπει να κοιτάω περισσότερο το χρονόμετρο, συμπαθάτε με. Φαντάζομαι θα έχετε την ευκαιρία να επανέλθετε. Ο Μπέντ Κόλμπερ. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Αξιότιμη προτινόμενη επίτροπε. Θα ήθελα να επανέλθω στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις και να τις συνδέσω. Η σα είπε ότι ανησυχεί τα 300 δις που εξήγηλε ως επενδύσεις ο κύριος Γιούνκερ ε, φοβάται ότι δεν θα υπάρξει ταχεία εφαρμογή. Εγώ φοβάμαι για το αντίθετο, ότι θα εφαρμοστούν γρήγορα χωρίς να υπάρξει προστιθέμενη αξία ε, που να είναι με τρόπο αηφόρο και βιώσιμο στη διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών. Ήδη έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις 220 ε, δις ε, και πληρωμές 143. Φοβάμαι ότι η Ένωση μπορεί να έχει και νομικά προβλήματα γιατί δεν επιτρέπεται να δανείζεται και να έχει χρέος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα πώς σκέφτεστε να το ξεπεράσετε, πώς θα κάνετε αυτό το σπαγκάτ για να συνδυάσετε και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Όλοι συμφωνούμε εδώ ότι πρέπει να γίνεται χρηστή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων και είναι μέρη μου αυτό. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο στόχος μας ποιος είναι να έχουμε αυτή τη φορά μικρότερα ποσά. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε περικοπεί 2,4% στην ανάληψη υποχρεώσεων και λίγο παραπάνω 2,7% δεν απαθώμε στις πληρωμές. Ε, λίγο λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν και όταν είναι υψηλότερες οι απαιτήσει και η απορρόφηση ε, χρειάζεται βελτίωση σε πολλές χώρες. Το πώς λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε και θα αξιοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι το 80% εκτελείται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Πώς όμως θα έχουμε πάντα ευθυγραμμισμένες τις προτεραιότητες με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά σίγουρα είναι ένα καθήκον που εγώ είμαι προσιλωμένη να συνεχίσω. Για τα 300 δις τώρα. Γιατί τα συζητούμε, για ποιο λόγο. Διότι αυτό που σήμερα αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη είναι ότι λεφτά υπάρχουν και πολλά στο σύστημα, στις τράπεζες, τα οποία κοιμούνται είναι τελείως αδρανή και θα πρέπει να ξυπνήσουμε αυτή την ενέργεια για τις επιχειρήσεις για να επενδύουν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες για να μπορεί να λειτουργήσει η μηχανή, το σύστημα ακόμα περισσότερο. Τα 300 δις βεβαίως είναι και για δημόσιες επενδύσεις και αντίστοιχα προγράμματα, αλλά για να ενισχύσουν, να τονώσουν την οικονομία για να δημιουργηθεί εργασία. Ας πούμε, στην ψηφιακή αγορά. Τεράστιες ε, ευκαιρίες που ακόμα δεν έχουμε αξιοποιήσει. Θα επανέλθετε, λέει ο πρόεδρος, μην ενισχύετε. Θα έχετε την ευκαιρία οπωσδήποτε. Ο Ζεράρ Ντεπρέ, παρακαλώ. Μάλιστα. Κυρία Επίτροπε. Διότι είστε ακόμα επίτροπος, αν δεν απατώμε. Καλώς ορίσατε εξ ονόματος της ομάδας μου και θα ήθελα να τονίσω ότι ε, η φήμη που σας συνοδεύει είναι πολύ ε, κολακευτική για τον τρόπο με τον οποίο ασκείτε τα καθήκοντά σας στην παρούσα θητεία. Εγώ όμως δεν έχω ικανοποιηθεί πλήρως από τις απαντήσεις ε, για τις πληρωμές. Ε, διάβασα την επιστολή που σας απίφθηνε ο κύριος Γιούνκερ και λέει η πρώτη σας ευθύνη είναι να καταρτήσετε ένα σχέδιο για τις προτεραιότητες για τις πληρωμές. Όποιος λέει προτεραιότητες εννοεί ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι δευτερεύοντα, άρα δεν θα πληρωθούν. Και είπατε λοιπόν εσείς ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός του 2014 και ο προϋπολογισμός του 2015 μας είπε ο Επίτροπος Ντομινίκ ότι αυτά αρκούν για να σταματήσει κατηφόρα. Η κατηφόρα οποία είναι διαρκή και μόνιμη τώρα. Και είτε στην ενδιάμεση αναθεώρηση, είτε το 2019 θα αλλάξετε τα πράγματα. Μα δεν θα έχουμε χρόνο κύριε Επιτροπέ, πήγουν αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα στρατηγικό σχέδιο, μπορείτε να υπολογίζετε στο Κοινοβούλιο για να το κάνει αυτό, αλλά θα πρέπει να απορροφηθεί το συντομότερο ε, αυτό το έλλειμμα των πληρωμών. Να λήξει αυτή η υπόθεση. Πώς θα γίνει θα συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν ε, θέλω να αποφύγω να απαντήσω, θα το τονίσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά με τη σειρά. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ευελιξία για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τις πληρωμές και να δώσουμε χώρο για αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό μας με τρόπο πιο παραγωγικό, χωρίς καθυστερήσεις και αναβολές. Εξού και η υπόσχεση του κυρίου Γιούνκερ για τα 300 δισεκατομμύρια. Τρεις μήνες έχουμε, δεσμευτήκαμε για να έρθουμε σε εσά και το Συμβούλιο και να πούμε ειδού πώς σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για επενδύσεις δεδομένων των περιορισμών ε, που σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό τώρα θα γίνει ε, και σε σχέση με τη συζήτηση για μεγαλύτερα στρατηγικά θέματα βεβαίω, α πούμε, οι ίδιοι πόροι είναι ένα τεράστιο θέμα, στρατηγικό, οπωσδήποτε πρέπει να το δούμε. Και να πούμε ότι ορίστε τώρα, είναι έτσι η κατανομή του προπολογισμού. Μα αυτή είναι γνωστή, 28 χώρε ε, σε διάφορου τομεί έχουμε συμφωνήσει τι πρέπει να γίνει, πάνω κάτω αυτά είναι ρυθμισμένα το περιθώριο ελιγμών είναι κάπως περιορισμένο. Αλλά ας το δούμε θετικά. Έχουμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα, πολύ περισσότερα για την ανταγωνιστικότητα, περισσότερα για τις ε, ζώντιες δράσεις και προγράμματα και για να μην έχουμε πρόβλημα αυτή τη φορά, θα σας πω ότι θα επανέλθω για αυτό το θέμα επανειλημμένα ξανά και ξανά, διότι είναι κρίσιμο για μας με τρόπο διαδραστικό να βοηθήσουμε την Ευρώπη να προχωρήσει. Ευχαριστούμε. Λιάτ Νιάντα. Ευχαριστώ πολύ. Όντω υποφέρουν από τη λιτότητα οι λαοί της Ευρώπης και στην Ιρλανδία έχουμε μια φόρητη κατάσταση και με τις ελευτικές κοινότητες, για παράδειγμα, να βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να βρούνε αρκετά χρήματα για να έχουν να τις οικογένειές τους. Εσείς είσαστε από τη Βουλγαρία και βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδυλιά. Εμείς έχουμε επίσης τεράστιο προβλήμα, πρόβλημα. Έχουμε 200 οι οποίοι μεταναστεύουν κάθε μέρα, πηγαίνουν σε άλλες χώρες και μάλιστα είναι και νέοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Τι εγγύσεις λοιπόν μπορείτε εσείς να μας δώσετε ότι θα καταφέρετε να πείσετε τις χώρες μέλη έγκαιρα να επενδύσουν στα, προγράμματα αυτά τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και τι αντιπροτάσεις έχετε για να αντιμετωπίσετε τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν ακόμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Θα εφαρμόσετε μέσα όπως είναι το κριτήριο της εξαίρεσης λόγω κρίσης. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που θέσατε το ζήτημα αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η μία πτυχή είναι ότι στην μεταπολεμική μας ιστορία για πρώτη φορά, για πρώτη φορά βλέπουμε σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές η φτώχεια να αυξάνεται, να μειώνεται. Και αυτό είναι βέβαια πολύ μεγάλη ανησυχία για όλους μας η αυτή. Γι' αυτό και στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κονδύλια που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της απασχόλησης νέων ευκαιριών, αλλά και το Κοινωνικό Ταμείο προσπαθεί να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους μεταξύ των συμπολιτών μας. Είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Είναι δημογραφικά τα δεδομένα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πληθυσμό στην Ευρώπη γυράσκει και ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι μορφωμένοι, ψάχνουν δουλειά εκτός Ευρώπης. Κάποιος έγραψε πρόσφατα είναι στη Γαλιφόρνια και αναρωτιέται θα υπάρχουν δουλειές για να γυρίσει πίσω στην Ευρώπη. Αν λοιπόν δεν επικεντρωθεί η Ευρώπη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, ιδιαίτερα στις νέες βιομηχανίες, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού, να παλύψουμε τη φτώχεια, να βοηθήσουμε τους συμπολίτε μας, να δώσουμε μια νέα όθηση σε αυτούς που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση θα δείτε ότι με τα 300 δισεκατομμύρια δεν μιλάμε μόνο για χρήματα, μιλάμε όμως και για πολιτικές, πώς θα έρθουν τα εμπόδια που δυσκολεύουν την ανάπτυξη να έρθει. Όντως, κάποιοι βρίσκονται πιο πίσω, δεν θα συμβαίνει αυτό όμως πάντα. Φυσικά και θέλω στον προϋπολογισμό κονδύλια τα οποία να βοηθούν τα προγράμματα αντιμετώπισης της κρίσης. Δεν έχω χρόνο, αλλά θα επανέλθω, να ξέρετε. σε ευχαριστούμε. Η Μόνικα Βάνα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Προτινόμενη Επίτροπε. Μιλήσατε για τις επιπτώσεις ε, του προϋπολογισμού της Ένωσης στη ζωή των πολιτών μας και πόσο σημαντική είναι η πολιτική ισότητα. Από πλευρά των Πρασίνων δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας και ρωτώ και το θέμα του φύλου έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Υπάρχει μια μελέτη από το έτος 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θέματα ισότητας και καταλήγει στο ανησυχητικό συμπέρασμα ότι βεβαίως υπάρχει το gender budgeting από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο, δηλαδή η συμπερίληψη του φύλου ε, στον προϋπολογισμό αλλά δεν εξασφαλίζει καθόλου την ισότητα ε, σε όλη τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτρα. Και ρωτώ, πώς θα εξασφαλίσετε με συγκεκριμένα βήματα ακριβώς την ε, ανάλυση του προπολογισμού με βάση το φύλλο, τι επιπτώσεις θα έχει σε άνδρες και γυναίκες. Και τώρα ε, ρωτώ για το έτος 2016 πλέον για την κατάρτιση εκείνου του προπολογισμού. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας αυτή. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν φροντίζει ολόκληρο τον πληθυσμό και τους άντρε και τις γυναίκες και το να λαμβάνουμε υπόψη μας τη διάσταση του φίλου στον προπολογισμό έχει να κάνει και με την παραγωγικότητα, έχει να κάνει με το να έχουμε την καλύτερη απόδοση των επενδύσεών μας. Στα σημερινά μου καθήκοντα και ναι, βεβαίως η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν ε, τιμή για μένα που το είχα σαν αρμοδιότητα. Και γίνανε τεράστιε προσπάθειες για να λαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές η διάσταση του φίλου υπόψη. Σε όλες μας τις δραστηριότητε. Δεν είναι εύκολο. Καταρτίζουμε ανθρώπους κλπ. Στα μελλοντικά μου καθήκοντα υπάρχουν προγράμματα όπου αυτό έχει ήδη γίνει. Στην επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε περισσότερα πράγματα εκεί που είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Πώς θα έχουμε κριτήρια για την ε, ισότητα παντού. Το κατά πόσο θα πετύχουμε ή όχι εξαρτάται από τις χώρες μέλη. 80% ε, των δικών μας κονδυλίων πηγαίνουν σε μεικτή διαχείριση. Το να έχεις νερό δεν φτάνει, δεν φτάνει μάλλον να πας, να πας και το άλογο να πιει. Συνεπώς, για μένα το βασικό καθήκον είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε τον προπολογισμό, ναι, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται, αλλά μετά πώς θα δημιουργηθεί αυτή η νοοτροπία, αυτή η κοινή κατανόηση για όλους, ότι δεν πρόκειται μόνο για άτομα, για γυναίκες, πρόκειται για την επίδοση της δικιάς μας οικονομίας πάνω απ' όλα. Μάρκο Ζάνι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρει ερωτήσει για τι τρεις προκλήσεις που έχετε κύριε Γεωργίου, κατά την θητεία σας αυτή πρώτα όλα, όσον αφορά τι πιστώσει πληρωμών για να επανέλθω στο ίδιο θέμα μας είπατε ακριβώς τι σκοπεύετε να κάνετε ούτω ώστε να μπορέσετε ε, να αντιμετωπίσετε αυτές τις εκκρεμούσες πληρωμές, να σταθεροποιήσετε την κατάσταση. Αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να ακούσουμε είναι τι διαρθρωτικού χαρακτήρα λύσεις έχετε κατά νου, ούτως ώστε να αποφύγουμε το πρόβλημα αυτό, να το αντιμετωπίσουμε και πάλι στο μέλλον. Να μην γίνει ό,τι έγινε στο παρελθόν, όπου κάθε χρόνο είχαμε ε, ανεξόφλητους λογαριασμούς, οι οποίοι ε, σωρεύονται. Οπότε ίσως ε, θα πρέπει κάποιες... Ε, πιστώσεις υποχρεώσεων να τις αναθεωρήσουμε και να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε την κατάσταση. Μία άλλη πρόκληση είναι το να έχουμε κάποιο είδου δραστικέ περικοπέ όσον αφορά τι διοικητικέ δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαράδεκτο ε, σε συγκυρία κρίση και τόσε ανεργίε να έχουμε τόσε δαπάνε. Επίσης, τι θα, θέλετε, πώς θα, θα τα ζητήματα των υπαλλήλων των ε, υπηρεσιών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει επίσης όσον αφορά την τριπλή έδρα του Κοινοβουλίου που κοστίζει τόσα εκατομμύρια κάθε χρόνο, Γεωργίου. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις υποχρεώσεων, πρώτα-πρώτα να σας πω κάτι σε γενικό επίπεδο ότι οι υποχρεώσεις υπάρχουν για συγκεκριμένο λόγο. Δεν υπάρχουν για να κάνουμε τον ταχυδακτηλουργό και να τις ε, ανακατεύουμε έτσι και αλλιώς ανάλογα με το πόσα έχουμε να καταβάλουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Γίνεται το ένα επί τη βάση του άλλου πληρώνουμε επί τη βάση των υποχρεώσεων και γι' αυτό και έχουμε δύσκολε διαπραγματεύσει και θα πρέπει να ε, εστιάσουμε προσοχή μα για το πώ θα εκτελέσουμε καλύτερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον προπολογισμό για του Ευρωπαίου. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον των ε, πιστώσεων πληρωμών, εμεί ξεκινήσαμε πάρα πολύ σοβαρά κάποιο είδου ε, οριζόντιου χαρακτήρα, εγκάρσιο χαρακτήρα, προγραμματισμό για να δούμε πώ θα γίνεται η εκτέλεση ε, εφαρμογή των προγραμμάτων και να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαχείριση σε σχέση με την εξυπηρέτηση των εξοφλητέων των, των οφειλών μας. Ε, και κατά τη γνώμη αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν μπορέσουμε το, στο μέλλον να τα καταφέρουμε έτσι ε, μέσα στο στενόχρονο διάγραμμα που έχουμε αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Να, ε, ήδη στην γενική διεύθυνση της οποίας προείσταμε, ήδη αυτό έχει φέρει αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα την διοίκηση. Νομίζω ότι η Παγκόσμια Τράπεζα ε, θεωρείται ένα όργανο πάρα πολύ εύρεθμα λειτουργούν, αλλά ήρθα εδώ στην Κομισιόν και εντυπωσιάστηκα επίση. Θα πρέπει να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, να τι περιγωγέ θα κάνουμε σε όλε τι γενικέ διευθύνσει, να έχουμε περισσότερη ευελιξία και να δούμε πώ θα οργανωθούμε. Έχουμε τώρα μια νέα δομή τη Επιτροπή που προ τα εκεί πηγαίνει. Και θεωρώ ότι αυτό θα αποδώσει καρπούς, ότι δηλαδή θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια εξοικονόμηση δαπανών ε, με το να έχουμε καλύτερη διαχείριση του προσωπικού. Αυτά θα ήθελα να σας πω κι άλλα, αλλά τελείωσε ο χρόνος μου. Ο κύριος Συναδεινός, παρακαλώ. Δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Κάποιος από τους μη εγγεγραμμένους θέλει να μιλήσει αντί του κύριου Συναδεινού. Όχι. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν ο γύρος των ερωτήσεων εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Και τώρα θα περάσουμε στις μονομένες ερωτήσεις και πρώτα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρώτος, ο κύριος Σαλά Δαμασού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, το είδαμε από την αρχή της συνεδρίασης, ο προϋπολογισμός της Ένωσης ουσιαστικά κηρύσσει πάυση πληρωμών και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινδυνεύει να μην έχει τα μέσα να χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητες της, γιατί οι μόνες πιστώσεις που διατίθενται αφαιρώνονται στην πληρωμή του παρελθόντος. Γνωρίζουμε το καθεστώς αυτό ε, ε, και που οφείλεται. Έγινε μια περίεργη και ε, υπόγεια αλλαγή δεν είναι ανεξάρτητη η πόρη χρηματοδότησης πλέον του προπολογισμού, αλλά εθνική και το Κοινοβούλιο τελικά συμφώνησε για το δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά είχε βάλει ως προτεραιότητα και ως προϋπόθεση την αλλαγή αυτού του συστήματος. Υπάρχει η Επιτροπή Μόντι και χαίρομαι που θα συμμετάσχετε κι εσείς κατά δήλωσή σας αυτή. Πώς ε, εξετάζετε το ρόλο σας της αρμόδιας επιτρόπου σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου, καθενός ε, και αφετέρου στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμασούρ και για τα όσα κάνατε ως πρόεδρος Επιτροπής αυτής για να βοηθήσετε ε, την ε, υπόθεση. Και στο παρελθόν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω πολύ να εργαστούμε σκληρά με όλη μας την ενέργεια και τις προτάσεις στην ομάδα υψηλού επίπεδου και να κάνουμε προτάσεις ακριβά αξιόπιστες. Γιατί τι είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια των ετών. Δεν μας βοηθάει ε, ο τρόπος με τον οποίο ε, καταρτίζει το προϋπολογισμός έχει μειωθεί το ποσοστό των ιδίων πόρων και έχει αυξηθεί το ποσοστό από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, από το ΕΠ. Και σε καιρούς οικονομικής στενότητας αυτό οδηγεί σε πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Και έρχονται οι φίλοι της ε, συνοχής απέναντι στους φίλους της Γεωργίας, οι καθαροί συνεισφορείς απέναντι στους καθαρούς αποδέκτες, το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Έρχονται διάφοροι αντιμέτωποι με διαφόρους άλλους. Αυτό δεν βοηθάει την ενότητα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο το θέμα ε, ε, λογιστικό πόθεν ε, βρισκόνται τα χρήματα, αλλά ο τρόπος που λειτουργούμε και πώς επηρεάζεται από τον προϋπολογισμό γενικότερα. Ελπίζω να κάνουμε προτάσεις οι οποίες θα είναι πολιτικά βιώσιμες και θα μπορέσουν τουλάχιστον να μας οδηγήσουν σε αλλαγή κατεύθυνσης. Γνωρίζουμε όλη την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτού. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην άποψή της. Ο δικός μου ρόλος θα είναι πάρα πολύ ε, πρωταγωνιστικός με ενεργή συμμετοχή και ο πρώτος αντιπρόεδρος θα συμμετέχει εκεί και άλλοι αντιπρόεδροι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε τμήμα της διαδικασίας. Με έκβαση που θα είναι πολιτικά αποφασιστική. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ Τωμά. Ευχαριστώ. Προτεραιότητα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι τα 300 δισεκατομμύρια για την απασχόληση και την ανάπτυξη. 25 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε συζητήθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας προκειμένου να γίνουν βιώσιμες επενδύσεις και να δοθεί όθηση στην απασχόληση. 20 με 40 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να πάνε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση αυτή και την εφαρμογή της. Πώς θα διασφαλίσουμε το δημοκρατικό έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων αυτών. Επίτα, αναφερθήκατε πριν στα ομόλογα έργου. Και ευχαριστώ τον Κόρον Φαμ για το μέχρι τώρα έργο του. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ιδιωτικούς επενδυτές να χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα υποδομών. Υπάρχουν όμως δυσκολίες. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος δεν θα είναι ο μόνος ο οποίος θα αναλάβει τον κίνδυνο των επενδύσεων αυτών, αν καταλήξουν σε κάποια αποτυχία, ενώ οι επενδυτές μόνο θα κερδίσουν αν πάει καλά το έργο. Και γρήγορα θέλω να ακούσω και τη γνώμη σας για την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού ταμείου θα μειωθούν οι διατάξεις των διαρθρωτικών ταμείων μηχανισμών που θα καταλήξουν έχουν τον Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μόνη τράπεζα επενδύσεων. Απάντηση. Πολύ καλές όλες αυτές οι ερωτήσεις σας. Πρώτον, δεν πρέπει να βιαζόμαστε για τα 300 δισεκατομμύρια. Γιατί, όπως είπαμε, το είπε ο νέος πρόεδρος, αλλά θα δουλέψει καλά το σύστημα αυτό μόνο εφόσον συνεργαστούμε καλά όλοι μεταξύ μας. Οπότε και εσείς θα μπορέσετε να μιλήσετε με τον πρόεδρο και εννοείται ότι σε τρεις μήνες θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες για το τι θα γίνει με το ποσό αυτό. Είμαστε σώμα επιτρόπων, λειτουργούμε ως ομάδα και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε. Δεύτερον, όσον αφορά τα καινοτόμα μέσα και τον έλεγχό τους, το δημοκρατικό τους έλεγχο. Συμφωνώ μαζί σας για το ότι δεν θα έπρεπε να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι και να αφήσουμε τους κινδύνους τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και τα κέρδη μόνο στους επενδυτές. Αλλά δεν είναι αυτό που προτείνουμε και δεν είναι αυτό που θα κάνουμε. Αυτό που προτείνουμε είναι να δούμε τους περιορισμούς που υπάρχουν και τις δυσκολίες έτσι ώστε να φτάσουν οι επενδύσεις, να κινηθούν και να έχουμε κάτι συγκεκριμένο για αυτού του είδους επενδύσεις. Δούλεψα στην Παγκόσμια Τράπεζα 17 χρόνια και μπορώ να σας πω ότι οι μηχανισμοί ελέγχου μπορεί να είναι πάρα πολύ ισχυρή για αυτού του είδους τις επενδύσεις, όπως είναι και για άλλες περιπτώσεις χρηματοδότησης. Μπορούμε λοιπόν κάλλιστα να διαχειριστούμε υπεύθυνα το δημόσιο χρήμα με την ευελιξία έτσι όπως προτείνεται αυτή σήμερα. Και μια που έχω ακόμα χρόνο. Πιστεύω ότι το θέμα ελέγχου των καινοτόμων αυτών μέσων χρηματοδότησης έχει πολύ μεγάλη σημασία και θεωρώ προνόμιο για μένα που θα μπορώ εφόσον επιβεβαιωθώ στο χαρτοφυλάκιό μου να αναλάβω αυτό το ζήτημα. Γιατί προσωπικά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι μπορεί να γίνει. Και πραγματικά δεσμεύομαι εγγυώμαι ότι δεν θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και θα σπαταλήσουμε τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Θα ήταν όμως από την άλλη σφάλμα να μην προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της μόχλευσης του χρήματος. Γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται να έχουμε περισσότερη καινοτομία, δημιουργικότητα και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει στις χώρες μας. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Είδατε το χρονόμετρο και τώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, στις γραπτές σας απαντήσεις ε, που δώσατε στις ερωτήσεις μας, οι οποίες κατά τα είναι εξαιρετικές και οφείλω να το πω, αναφερθήκατε και στο εξή. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μεταξύ έχουν πρόβλημα αξιοπιστίας οι οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χαίρουν και τεράστια σε και εκτίμησης στα μάτια των πολιτών στην Ένωση. Πώς βελτιώνεται αυτό. Ένα βήμα είναι με περισσότερη διαφάνεια. Θα πρέπει να καταλάβουν και πάλι οι πολίτες για ποιο λόγο υπάρχουν τα θεσμικά όργανα και γιατί κοστίζουν τόσα πολλά χρήματα. Και έχω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Το 1990 είχαμε τρεις οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, agencies. Από το 2004 ε, ε, άρχισαν να διπλασιάζονται και τώρα έχουμε περίπου 40. Μα χρειάζονται όλοι αυτοί, ορισμένοι δρεύουν και στις Βρυξέλλες. Πρέπει να έχουμε τόσους πολλούς ε, οργανισμούς. Θα φροντίσετε να υπάρξει αξιολόγηση για το πόσο έχουν αξία και μας χρειάζονται όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. πολύ. Μπορώ να σας πω για την διαφάνεια. Συμφωνώ. 100% για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα, η διαφάνεια είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουν τα χρήματά μας από λαθροχειρίες ακόμα και σε ένα περιβάλλον διαφθοράς όπου υπάρχει διαφάνεια υπάρχουν αποτελέσματα. Είχαμε και στην προηγούμενη μου ε, σταδιοδρομία. Είχα πάει στο Ταταρστάν, στην Ινδονησία και εκεί όποτε εφαρμόσαμε την διαφάνεια και ζητήσαμε να μας πούνε τι ακριβώς έγινε με τις δαπάνες, ε, τότε οι κοινότητες συγκρότησαν ένα σύστημα ελέγχου. Γι' αυτό σας λέω ότι αποδίδει αυτή η λύση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλη διαφάνεια, αλλά θα πρέπει να είναι και φιλικό στο χρήστη το σύστημα. Πολλές φορές θέλει κανείς κάτι να μάθει και ψάχνει και ψάχνει για τη δουλειά μας και δεν βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Και όμως οι πληροφορίες κάπου βρίσκονται. Και επίσης αυτό είναι το τμήμα της αποστολής μου. Το πώς η διαφάνεια θα λειτουργήσει όσο πιο φιλικά γίνεται για το χρήστη. Τώρα όσον αφορά τους οργανισμούς και υπηρεσίες, η κάθε μία και κάθε οργανισμός φτιάχνει και κάποιο λόγο για να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ε, συγκεκριμένο. Υγεία και προστασία της. Ή για σκοπούς ε, έρευνας, ε, καινοτομία κλπ. Όντως, σας ομολογώ ότι θα πρέπει να μάθω περισσότερο για τον κόσμο των υπηρεσιών και οργανισμών της κοινότητας. Αλλά γενικώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν κάποιος θέλει αποτελεσματική χρήση των πόρων, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό διαφάνει. Κάτζα Κελάς. Μοιρές Αγελάδες. Είπε κύριε Γεωργίδα. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κάλλας. Σε Madame Amélie Jatenmaki qui la remplace. Okay. Merci. Αντικαθιστά όμως ε, τον κύριο Κάλλας, κύριε Γιατενμάκη. Στα φινλανδικά θα σας μιλήσω, λέει κύριε Άλλη. Στην τελευταία σας θητεία, κύριε Επίτροπε, τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Υπήρξατε εξαιρετικέ ικανότητε. Τώρα όμω το να λάβετε ένα όλο διαφορετικό χαρτοφυλάκιο. Και σας ερωτώ. Γιατί θεωρείτε ότι για το χαρτοφυλάκιο του προπολογισμού ο πιο ικανός, ο κατάλληλος άνθρωπος είστε εσείς, Γεργίβα. Και εγώ νομίζω ότι ο κύριος Γιούγκερ είναι ο πιο αρμόδιος να ρωτήσει αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Αλλά καλά, να σας πω γιατί θεωρώ ότι επελέγει. Ναι, είναι τεράστια η ευθύνη. Όντως, η πρώτη μου αντίδραση όταν το έμαθα, ε, τι να σου πω, ήταν ότι ανατρίχιαζα, δεν πειράζει είναι κομμένα κοντά τα μαλλιά μου, ήταν τόσο σοβαρό. Όμως, όμως, να να μιλήσουμε σοβαρά, κατάλαβα, κατέληξα στο ότι ο κύριος Γιούνκερ έχει κάποιο λόγο για να με επιλέξει. Για δύο λόγους συγκεκριμένα. Γιατί επαγγελματικά έχω ασχοληθεί με χρήματα, με κεφάλαια. Ήμουν ε, ε, στο, στο Προεδρείο της Παγκόσμιας Τράπεζας, συγκεκριμένα στο γραφείο του Αντιπρόεδρου. Ασχολήθηκα με όλα τα τμήματα της Παγκόσμιας Τράπεζας σε εκείνο το επίπεδο και θεώρησα ότι έχω τέτοιες ευθύνες ε, σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά και νομίζω ότι οι επιδόσεις μου ήταν αξιόλογες. Επίσης, ο δεύτερος λόγος που επελέγει είναι ο εξή. Νομίζω ότι απέδειξα την ανεξαρτησία μου για το ότι δεν δέχομαι εντολές από κανέναν και ότι γνώμονας μου είναι μόνο το συμφέρον των Ευρωπαίων. Και αυτό νομίζω ότι είναι η βασική προϋπόθεση για να λάβει κανείς αυτό το πόστο. Και επίσης ότι δουλεύω σκληρά. Ε, θα βοηθήσει και αυτό. Κυρία Λιάντ Μυριάντα, μιλάμε για δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια μίλια βέβαια μακριά από αυτούς οι οποίοι υποφέρουν από τη φτώχεια. Ξέρουμε ότι ένα παιδί στα πέντε ζει στη φτώχεια στην Ιρλανδία, για παράδειγμα. Και ξέρετε κι εσείς κι εγώ ότι οι πόροι οι οποίοι δίνονται στα προγράμματα όπως εγγύηση για την νεολαία κτλ. δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των πραγματικών επενδύσεων σε βιώσιμη επαργωγή και ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών κινδυλίων μέσω των λεγόμενων καινοτόμων οικονομικών μέσων και προγραμμάτων χρειάζονται βιώσιμες λύσεις. Αυτό το οποίο δημιούργησε την οικονομική κρίση ήταν ακριβώς η χρήση κερδοσκοπικών μέσων. Εδώ χρειαζόμαστε μια προοδευτική κοινωνική Ευρώπη. Δεδομένης της ιστορίας μας λοιπόν, πιστεύετε ότι κερδοσκοπικά μέσα είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Απάντηση. Δεδομένου του παρόντος και των προοπτικών που έχουμε για το μέλλον, πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους Ευρωπαίους αν δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες εδώ στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ελευθερώσουμε το δυναμικό που έχουν οι επιχειρηματίες μας και ιδιαίτερα οι νέοι επιχειρηματίες μας. Προς το παρόν, δεν βλέπουμε αρκετή όθηση επενδύσεων στην Ευρώπη. Δεν βλέπουμε αρκετή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και εμείς έχουμε την ευθύνη να παίξουμε τον ρόλο μας και εμείς επ' αυτού. Μην ξεχνάμε ότι τα καινοτόμα οικονομικά μέσα αποτελούν ένα μικρό μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, 9 δισεκατομμύρια, το τριπλό, αλλά ξεκινώντας από πολύ πιο χαμηλή βάση. Και για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την αξιολόγηση της εμπειρίας από διάφορες πρωτοβουλίες που θα έχουν γίνει, ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να έχουμε το θάρρος. Και αν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, πρέπει να το ακυρώσουμε, δεν πρέπει να το επεκτείνουμε περισσότερο. Τα πειραματικά προγράμματα και αυτό ακριβώς υπάρχουν. Αν πάνε καλά, έχει καλός. Αν δεν πάνε καλά, ας πεθάνουν. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά ενθουσιώδεις να προχωρήσουμε αν προηγουμένως δεν έχει γίνει μια αξιολόγηση και θα γίνει. Αυτό σας το υπόσχομαι. Συγχρόνως βέβαια πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τους πιο ευάλωτους, για αυτούς που υποφέρουν περισσότερο, που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η εγγύηση για την νεολαία είναι σημαντικό. Έχουμε 6 δισεκατομμύρια και ελπίζω να είμαι η Επίτροπος η οποία θα αυξήσει το ποσό αυτό και θα επεκτείνει τη δράση του προγράμματος. Πρόεδρος, Ιντρακ Ευχαριστώ κυρία Κεωργίευα. Θέλω συγχαρώ το βουλγαρικό λαό καταρχάς που αντίθετα με άλλους ε, λαούς ε, διόρισε κάποιον ως επίτροπο ανεξάρτητο από την πολιτική, μακριά από την πολιτική, που ξέρει τι εστί ε, η πραγματική ζωή και έχει και περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Γι' αυτό εμείς οι πράσινοι σας υποστηρίζουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένα θέμα που επήγει. Ε, το 20% του πολιετές του πλαισίου ε, δεν επαρκεί για το περιβάλλον. Πώς προτίθεστε λοιπόν να αξιοποιήσετε τις γνώσεις σας που έχετε για τα περιβαλλοντικά θέματα ε, για να καταπολεμήσουμε την κρίση του περιβάλλοντος περισσότερο και με περισσότερο πρασίνισμα του προπολογισμού. Και στη Γεωργία και ε, παντού να εντάσσετε και το περιβάλλον ε, έτσι ώστε να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή γιατί μια στεναρή και ισχυρή πολιτική δεν αρκεί να εξαντλείται στις δηλώσεις και στις προβλέψεις και στις εξαγγελίες και στις προθέσεις. Ευχαριστώ πολύ ε, που αναφερθήκατε στους πολλαπλούς στόχους του προϋπολογισμού. Πάντα στη δράση μας, σε οτιδήποτε κάνουμε, θα πρέπει να φιλοδοξούμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και από την προηγούμενη μου εμπειρία, την περιβαλλοντική και την επαγγελματική, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω διαπιστώσει ότι η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός. Και ε, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι υπαριθμόν ένα αγώνας που θα κληθούμε να δώσουμε. Για φέτος, όπως γνωρίζετε, είμαστε στο 12,5% από το 20% που θέλαμε να αφιερώσουμε σε αυτό το σκοπό. Ε, και η φιλοδοξία μου είναι να φτάσουμε στο 20 και μάλιστα εγώ θα χαιρόμουν αν το ξεπερνούσαμε κιόλα. Ε, ε, ε, έχουν αρχίσει κάποια προγράμματα να εφαρμόζονται, αλλά θα αποδώσουν το 2016 μόνο. Ενώ ταυτόχρονα ε, στη γεωργική πολιτική προχωρούν και προς το λεγόμενο πρασίνισμα και στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Όταν προετοιμαζόμουν για την ακρόαση, διάβαζα τόμους εγγράφων και βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. 138.000 βιολογικοί καλλιεργητές ήδη ε, υποφελούνται από το πρόγραμμα ε, και για πιο υγιεινά τρόφιμα αλλά και για καλύτερη νοοτροπία ως προς την πράσινη οικονομία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται στον προϋπολογισμό και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό, τι κάνουμε με τα χρήματα για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά τι κάνουμε και με τα κτίρια. Στην καθημερινή μας δουλειά πώς αντιμετωπίζουμε αυτό τον κίνδυνο και την απειλή της κλιματικής αλλαγής. Jonathan Arnott. You told us that you are... Μας είπατε ότι θα θέλατε πάρα πολύ να έχει μία και μόνη έδρα κοινοβούλιο το είπατε σχετικά του συναδέλφου. Για πετε μα, είναι πάρα πολύ φορολογούμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ιταλία, που θεωρούν ότι το να πηγαίνουν έρχεται το κοινοβούλιο κάθε μήνα του Βρυξέλλε στο Στρασβούργο και να καταβάλλονται γι' αυτό εκατοντάδε ε, εκατομμύρια κάθε μήνα, ε, σημαίνει ότι, ότι έχει χρήματα ο προπολογισμό. Ε, και έτσι διασπαθούν τα χρήματα. Για πέστε μας, εσείς τι θα κάνετε. Πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα. Θα θέλατε να υπάρχει μόνο, μόνο μία έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι να κάνετε εξοικονόμηση. Πώς θα μπορείτε να έχετε κάποιο είδους ε, κριτήρια που να προϋπάρχουν για όλα τα προγράμματα και έργα της κοινότητας και να ξέρουμε αν πετύχανε ή απέτυχαν. Γιατί θα πρέπει να δούμε ε, το ότι όλο ένα και περισσότερο προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι. Όλο ένα και περισσότερο μεγαλώνει αυτός ο στρατός των Ευρωπαίων Γραφειοκρατών που καταλήγει πιο μεγάλος από τον Βρετανικό στρατό. I'm getting worried about the size of the British Army. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ γι' αυτό και ανησυχώ για το μέγεθος του Βρετανικού στρατού, λέει η κυρία Γεωργίου. Για την πρώτη σας ερώτηση. Με κάθε σεβασμό θα σας πω το εξής. Γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο είπατε απαιτεί τροποποίηση των συνθήκων. Κάποιοι συνάδελφοι ε, που ασχολούνται με τα με, με, με τα θέματα τη ανθρωπιστική βοηθείας λένε ότι κάνω θαύματα στη δουλειά μου. Ε, όχι, δεν μπορώ να κάνω θαύματα σε αυτό. Είναι θέμα των συνθήκων. Αρμόδιοι αυτοί μπορούν να τροποποιήσουν τη συνθήκη. Τώρα όσον αφορά το πώ θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, στο τι ξοδεύουμε, Ακριβώ αυτό σημαίνει αποτελεσματικό προπολογισμό. Και εμεί αυτό θέλουμε και να κάνουμε με ένα νέο ε, δημιουργικό πολιτές πλαίσιο και ακριβώς και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να μας υποπτεύει, να συνεργάζεται μαζί μας όπως και κάνει. Αλλά δεν είναι κάτι το εύκολο γιατί όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση του προπολογισμού θα πρέπει κανείς ε, να καταρτίζοντας τον προπολογισμό όχι μόνο να προβλέψει ε, το πόσα θα δαπανίσει αλλά και ποιες θα είναι επιπτώσεις από αυτά που δαπανώνται και το μεγάλο αιώνιο πρόβλημα είναι το ότι πάρα πολύ συχνά αυτό αυτό, αυτός ο λόγος μας πρόχνει στο να προσέχουμε αυτά που μετρώνται εύκολα και όχι να προσέχουμε αυτά που είναι τα πιο σημαντικά. Οπότε για να είμαστε αποδοτικοί οδηγούμεθα σε κάποιο είδους ε, αθέλητες αρνητικές συνέπειες. Άρα θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να προχωρήσει κανείς πάντως δικαιολογία δεν υπάρχει καμία όσον αφορά αυτό το οποίο ερωτήσατε που είμαι σίγουρος ότι και άλλοι θα ήθελαν να ρωτήσουν. Οπότε και ειλικρινά σας ε, υπόσχομαι να ασχοληθώ ακριβώς με αυτό το θέμα. Ε, ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Στεβάν Κονζάλης Μπόνς. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφια, ε, Επίτροπε, οι Ευρωπαίοι πολίτες όλο και πιο πολύ αναρωτιούνται αν κάνει καλά πράγματα η Ευρώπη. Έλεγα λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες να όλο και πιο πολύ κατά πόσο είναι καλό να έχουμε την Ευρώπη, ευρωσκεπτικισμός δηλαδή, και πώς θα αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση ή το εμπάργο της Ρωσίας στα αγροτικά μας προϊόντα. Ο προπολογισμό είναι πολιτικό θέμα, αλλά ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν έχει αρκετή φιλοδοξία. Οι επικεφαλής της Ευρώπης δεν καταφέρνουν να φτάσουν ούτε στο 1% του ευρωπαϊκού πλούτου. Σας ρωτάω λοιπόν, εσείς είσαστε σε θέση να πείσετε τα μέλη του Συμβουλίου ότι μια μικρή αύξηση του προϋπολογισμού που είναι περιθωριακή για τα ταμεία τους θα είχε ιδιαίτερα θετικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή, με άλλα λόγια, συμφωνείτε ότι με λιγότερα χρήματα είναι αδύνατον να φτιάξουμε περισσότερη Ευρώπη. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι θλιβερό ότι στο τέλος των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η απόφαση ήταν ένα μικρό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα έχουμε αυτό που έχουμε. Και νομίζω ότι είναι περισσότερο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή αυτού που έχουμε και να δείξουμε την αξία των δράσεών μας. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όσοι αγαπούν την Ευρώπη πρέπει όντως να ανησυχούν για το γεγονός ότι χάνουν οι Ευρωπαίοι την εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε φυσικά να συζητήσουμε για τις αιτίε, ποιο φταίει, ποιο έχει την ευθύνη κλπ. κλπ. Αλλά εγώ θα αναφερθώ μόνο στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Πρέπει λοιπόν εμείς να πούμε προς τα έξω και το τι κάνουμε. Πριν από λίγες μέρες ήμουν με έναν ευρωβουλευτή και τον ρώτησα, του είπα, ξέρετε ότι στη δικιά μου την πρωτεύουσα, στην πόλη όπου γεννήθηκα εγώ, έχουμε μετρό χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μπορούν πιο εύκολα να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους, οι επιχειρήσεις πιο εύκολα συναλλάζονται, υπάρχει περισσότερη ευημερία χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές τις ιστορίες όμως δεν τις λέμε προς τα έξω. Δεν τις λέμε αρκετά. Γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Όταν άρχισα πριν από λίγα χρόνια στην Επιτροπή, εγώ επέμενα για την προβολή των έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες. Και είχα πολλές αντιστάσεις, γιατί μου λέγανε «Μα όχι, δεν πρέπει, δεν έτσι, δεν αλλιώς». Όχι, και αυτό πρέπει να το κάνουμε, να προβάλλουμε το έργο μας. Γιατί να μην ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουμε και άμα δεν ξέρουν γιατί να μας στηρίξουν. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτό το θέμα το παίρνω πολύ στα σοβαρά. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Επικεντρωνόμαστε στις δαπάνες των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ξοδεύουμε σωστά τα χρήματά μας χωρίς απάτες και καταχρήσεις. Όμως όπως λέτε στις γραπτές σας απαντήσεις πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο και στα αποτελέσματα από τη χρήση των κονδυλίων. Γι' αυτό στο μέλλον πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα κατά πόσο τα ευρωπαϊκά κονδύλια έτσι όπως χρησιμοποιούνται πετυχαίνουν τους στόχους μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τα κοινοτικά κονδύλια και για τα 300 δισεκατομμύρια που προτείνει ο κύριος Γιούγκερ. Συνεπώς, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα ελέγξουμε τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και θα ελέγξουμε και την αποτελεσματικότητα, την απόδοση των, της χρήσης των κονδυλίων αυτών σε σχέση με τους στόχους μας, δηλαδή την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και έρχομαι τώρα στις οικονομικές μας εκκρεμότητες. Υπάρχει πρόβλημα με τις πληρωμές. Γιατί όμως δεν υπάρχει λύση, γιατί δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο. Είναι θέμα πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο λοιπόν. Οπότε ρωτάω, θα πείσετε το Συμβούλιο να υιοθετήσει διαφορετική θέση όσον αφορά τις πληρωμές, ώστε να μην έχουμε πια του λογαριασμούς. Απάντηση. Ναι, είναι αλήθεια ότι η ισορροπία αυτή ανάμεσα στην ε, καλύτερη χρήση των κονδυλίων και του ελέγχου είναι κάτι που πάντα μας απασχολεί, σίγουρα υπάρχουν εντάσεις, αλλά εγώ πιστεύω ότι η έλεγχη είναι αναγκαία. Αλλιώς, γιατί να μας εμπιστευτεί τα χρήματά του Ευρωπαίος Φορολογούμενος. Αλλά βέβαια ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο είναι να έχουμε φύση συστήματα όπου να υπάρχει κίνητρο εντοπισμού των σφαλμάτων, να έχουμε ανθρώπους που είναι καλά καταρτισμένοι για τον έλεγχο αυτό. Τα λόγια πρέπει να επικεντρωθούμε στη στήριξη και συγχρόνως να έχουμε πολύ δυνατά συστήματα ελέγχου. Ανα πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι στραβό με τον προπολογισμό μας, μα άμα συμβεί αυτό, τότε μας πάει πίσω, πολύ πίσω και αυτό είναι απαράδεκτο. Μηδέν ανοχή για την απάτη δεν είναι απλώς λόγια, δεν είναι σλόγγαν, είναι ανάγκη. Αν υπήρχε και μικρότερο νούμερο από το μηδέν θα έλεγα αυτό το νούμερο. Γιατί είναι ανάγκη να μην υπάρχουν ε, καταχρήσεις. Πρέπει όμως να μειωθεί και το κόστος των ελέγχων και ο καλύτερος τρόπος είναι ο καθένας από εμά να ενστερνιστεί την οτροπία αυτή αποτελεσμάτων και όχι να πούμε να αυτοί θα είναι οι ελεγκτές, αυτοί θα είναι οι σχεδιαστές των προγραμμάτων μας κλπ. Όχι, ο στόχος πρέπει να είναι κοινό για όλους. Και είναι εφικτό αυτό. Όσον αφορά το Συμβούλιο τώρα. Εγώ πιστεύω στο διάλογο, στις συνομιλίες και θέλω στο Συμβούλιο να δείξω ότι υπάρχει αξιοπιστία εδώ. Και αυτό θα κάνω. Θα τους προτείνω κάτι αξιόπιστο. Ίσως κάποια άλλη στιγμή να μπορέσω να τελειώσω την απάντησή μου. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Μπέρτ Κόλμεν. Ναι, κυρία πίτροπε. Τώρα μιλήσαμε πάρα πολύ για τις δαπάνες. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τα έσοδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασιζόταν στο παρελθόν σε ιδίους πόρους και αρκετά αξιόλογους και συνεισφορείς των κρατών μελών. Με την κατάργηση των τελωνιακών δασμών και εμποδίων μειώνονται όλο και περισσότερα οι ίδιοι πόροι. Οπότε αυξάνονται οι κρατικές συνεισφορές. Μοιραία. Τώρα, έχουμε τους καθαρούς συνεισφορείς, τους λεγόμενους και τους καθαρούς αποδέκτες. Ε, οι καθαροί αποδέκτες δεν παίρνουν το σύνολο πίσω. Μία χώρα που έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά παίρνει ένα κλάσμα πίσω. Δεν μπορεί να αλλάξει το σύστημα και να πληρώνονται λιγότερα χρήματα. Ε, έχουμε έτσι και εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραίο θα ήταν κάτι τέτοιο, θαυμάσιο οτιδήποτε θα μπορούσε να πλουστεύσει τον προπολογισμό μας. Ε, θα ήταν ευπρόσδεκτο γιατί έχει γίνει πάρα πολύ περίπλοκος και από την πλευρά των εσόδων και από την πλευρά των δαπανών και της διαχείρισης και της εκτέλεσης. Θα επανέλθω στους ιδίους πόρους για τους πόρους των εσόδων. Ο τρόπος με τον οποίο τώρα προσπαθούμε να αυξήσουμε τα έσοδα συμβάλλει στις συγκρούσεις και στις εντάσεις όπως είπατε και εσείς, ε, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε την αξία του ευρωπαϊκού προπολογισμού για τους πολίτες μας. Συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ζουν στις χώρες οι οποίες είναι καθαροί συνεισφορείς. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστό πόσο εποφελούνται εκείνοι από τον κοινοτικό προπολογισμό. Γιατί δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να αποτιμούμε και να μετρούμε πόσα χρήματα επιστρέφονται σε εταιρείες χωρών που είναι καθαροί συνεισφορείς και δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις σε χώρες της συνοχής και αποφελούνται από τα κοινοτικά κονδύλια. Έτσι πρέπει να ε, χτίζουμε γέφυρες εμείς αντί να διχάζουμε τις χώρες. Και η απλούστατη γέφυρα θα ήταν να φύγει όλο αυτό το επίμαχο θέμα. Χρειάζονται τέσσερις μέρες εργασίας των Ευρωπαίων για να φτιάξουν τον προπολογισμό. Πολύ καλύτερο θα ήταν να μειωθεί αυτός ο χρόνος. Εγώ είμαι ρεαλίστρια. Είναι δεδομένο αυτό το περιβάλλον, ε, σε αυτό θα εστιασώ για να μπορέσουμε να λειτουργούμε καλύτερα έτσι και με τους ίδιους πόρους σε ένα ενδεχόμενο διαφορετικό περιβάλλον. Ο Μιχαήλ Τόιρερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Στον προϋπολογισμό μας έχουμε την εξής κατάσταση. 81% είναι στις ε, συντρέχουσες μεικτές ε, αρμοδιότητες και τα διαχειρίζουν τα κράτη-μέλη. Και πάντα γίνονται συζητήσεις για την ποιότητα αυτής της διαχείρισης και την πολιτική αιρεσιμότητα, πόσο δεσμεύονται. Ας πούμε, οι εθνικές δηλώσεις διαχείρισης θα υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να εκτελούν καλύτερα το προπολογισμό. Γιατί παραμένει ε, μια κλασική λογική διαχείριση του προπολογισμού με λογιστικό τρόπο. Ε, μήπως θα πρέπει όμως να περάσουμε σε έναν προϋπολογισμό που να προσανατολίζεται στα πεπραγμένα και στις δραστηριότητες και στις επιδόσεις, performance-based budgeting. Και τι θέλετε να κάνετε για να βελτιώσετε και να μεταρρυθμίσετε τη δήλωση αξιοπιστίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Βεβαίω και θα υπάρχουν ε, και μου αρέσει το σύστημα αυτών των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας γιατί πολύ πολύ κακό το τελικά το έχουν σπαστεί το σύστημα πάρα πολύ για κράτη-μέλη 4-5 και μάλιστα ε, να δούμε τι θα γίνει με τις χώρες που έχουν κάποια προβλήματα με προπολογισμό και με εκτέλεση προγραμμάτων. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επεξεργαστεί μια πρόταση γι' αυτό και το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς θα πείσουμε τα κράτη-μέλη το ότι πρόκειται για πολύ εξαιρετική ιδέα. Να δούμε όμως γιατί υπάρχουν για κάποια κράτη-μέλη και κάποιες νομικές περιπλοκέ για να το πράξουν κάτι τέτοιο. Γιατί ε, να δούμε τι θα κάνουμε με τα κράτη που έχουν ομοσπονδιακή δομή. Αλλά όμως νομίζω ότι αυτό είναι ένας θετικός τρόπος να μπορέσουμε να εμπλακούμε περισσότερο, να εμπλέξουμε τα εθνικά κοινοβούλια να ασχοληθούν σε σχέση με την μη απορρόφηση κλπ. λοιπά... με τα προβλήματα τους πάντων με τους κοινωτικούς πόρους. Δεν είμαι τώρα τόσο σίγουρη για το ότι έχουμε βρει τον άριστο τρόπο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Γιατί ακόμα μέσα στη φάση κατά την οποία η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσεις δεν δουλεύουν σαν ομάδα για ένα στόχο. Μας θεωρούν κάτι σαν το, το φόβητρο. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στα αποτελέσματα. Τότε τα πάει καλύτερα. 100% θέλω να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να έχουμε κάποια προσοχή, να κάνουμε δηλαδή πρώτα πρώτο ό,τι είναι πιο εύκολο και προχωράμε προοδευτικά. We are aware of the work that out. Ε, ασχοληθήκατε με την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, ανταπόκριση στις κρίσεις και επομένω τώρα, εκτός από τις επιστώσεις υποχρεώσεων, ε, θέλω να ασχοληθείτε με κάποια άλλα θέματα με αυτά που γίνεται τώρα στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Μαλί, τη Συρία την Παλαιστίνη. Θα πρέπει να αυξηθεί η αρρωγή προς αυτές τις χώρες. Γιατί ουσιαστικά το ότι δίνουμε λιγότερο από το 2013 και τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν δημογραφικό πρόβλημα. Τι θα γίνει, η Frontex θα κάνει τίποτα για αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν στη Λαμπεντούσα, στις ακτές. Να έχουμε διεθνή συνεργασία για το άσυλο, την μετανάστευση, να σταματήσουν αυτές οι άθλιες περικοπές. Δεν θέλουμε ο κόσμος να γίνει έτσι που να μην θέλουμε να, να, βλέπουμε το πώς ζουν τα παιδιά σας ή τα παιδιά μας. Τι θα κάνετε επομένω για την οικοδόμηση κάποιας ειρήνης εκεί που χρειάζεται. Πάρα πολύ δύσκολο να σας απαντήσω δύο λεπτά, αλλά θα προσπαθήσω γιατί βεβαίως και με καίει αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε πρώτα-πρώτα για τη Frontex αλλά και την αναπτυξιακή βοήθεια. Βαθιά μου πεποίθηση είναι αυτό το οποίο και εάν ε, εγκρίνεται τον διορισμό μου θα το συνεχίσω είναι το ότι θα ήταν λάθος να προσεγγίσουμε τη μετανάστευση μόνο εστιάζοντας την προσοχή μας ε, μόνο στο από πού προέρχεται. Χρειάζεται τρίπλη προσέγγιση. Πρώτα-πρώτα προσέγγιση από τις ίδιες τις χώρες προέλευσης. Γιατί αυτοί ε, είναι τόσο απελπισμένοι, γιατί θέλουν να πάνε να σε σχεδίες και σκάφη ερήπια και να σκυλοπνίγονται. Επομένως χρειάζεται να υπάρχει ε, αναπτυξιακή βοήθεια για να εκκριζώσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Και που ξεκινάει δεύτερον, όσον αφορά τα δίκτυα των λαθρεμπόρων και δουλεμπόρων, χρειάζεται πάρα πολύ έντονη, εντατική παγκόσμια ε, συνεργασία. Οπότε και μετά να δούμε τι θα κάνουμε άπαξ και φτάνουν οι μετανάστες εδώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει βαθιά μέσα από την καρδιά μας να θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι η πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων θα πρέπει να αποτελέσει πολιτική μας αιμονία και σε σχέση με τους αμπισιακούς πόρους. Γιατί ακριβώς ξέρω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, το, το δούλεψε αυτό με την ανθρωπιστική βοήθεια. Πάρα πολύ εύθραστος ο, ο κόσμος. Ε, έχουμε και την κλιματική μεταβολή αλλά και τον εξτρεμισμό. Και μέσα σε αυτόν τον εύθραυστο κόσμο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο τραγωδίες εις βάρος κάποιων αθώων, αλλά βλέπουμε την αποτύπωση του, του, του, του πόσο βασανίζονται, πόσο υποφέρουν. Και αυτό για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ακριβώ ε, αυτή η αποτύπωση, αυτή η εντύπωση ε, του πόσο υποφέρει αυτός ο κόσμος έχει κάποιες συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές και άμεσες πάνω σε μας. Άρνοτ. Κύριε Επίτροπε, μας μιλήσατε για την πόλη σας ε, στη Βουλγαρία και το μετρό που φτιάχθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ένα παράδειγμα γιατί οι πολίτες πρέπει να είναι περισσότερο υπέρ Ευρώπης. Μα ο λόγος για τον οποίο χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη οι πολίτες είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί ξέρουν ότι είναι δικά τους τα χρήματα τα οποία στέλνονται στις Βρυξέλλες και μετά οι Βρυξέλλες έχει τα μπράβο. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Το ότι επικεντρώνει όλη την εξουσία στα χέρια της ε, η Ευρώπη εδώ στις Βρυξέλλες είναι ένα από τα προβλήματα. Οπότε η ερώτησή μου είναι αυτή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τομέα ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν χρησιμοποιηθεί και όπου τα κονδύλια δόθηκαν στις τοπικές αρχές ώστε να μπορέσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια να τα διαχειριστούν οι τοπικές αρχές για τις τοπικές τους ανάγκες. Απάντηση το μετρό έχει στη Σόφια μια στάση που ονομάζεται Ευρώπη, δεν ονομάζεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όντω είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες που έκαναν δυνατό αυτό το έργο. Για το θέμα τώρα του πού πρέπει να βρίσκεται η εξουσία. Εγώ πιστεύω ότι η εξουσία πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που μπορεί επιτυχώς να εκτελέσει ένα έργο. Και μερικές φορές δεν υπάρχει περιθώριο ούτε καν για την εθνική κυβέρνηση, πόσο μάλλον για την τοπική. Αλλά αλλού συμβαίνει το ανάποδο. Όταν μιλάμε για την έρευνα, με τη δικτύωση των πανεπιστημίων, τι κάνουμε. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να ανταγωνιστούμε τους μεγάλους γίγαντες, την Κίνα, την Ινδία. Και ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο από μόνο του θα δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα στον ανταγωνισμό αυτόν. Ενώ όλοι μαζί είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Θα έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά επίτροπο για την καλύτερη νομοθετική ρύθμιση. Και ακούω να λέτε από εσά ότι ναι το κάνουμε αλλά δεν έχει νόημα να γίνεται έτσι όπως γίνεται. Μα ήδη τα αξιολογούμε αυτά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο σκοπεύει να μας απαλλάξει από τα πράγματα τα οποία είτε είναι περιτά πια, είτε δεν χρειάζονται, είτε η αρχή της επικουρικότητας λέει ότι θα έπρεπε καλύτερα να είχαν γίνει σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα REFIT. Εγώ θα είμαι επίτροπος και για την προστασία του πολίτη. Και έχουμε συζητήσει για το θέμα της ε, της πολιτικής προστασίας. Ρόλος μας είναι να μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Σύγκριτ Μουρεσάν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε ε, για τα όσα είπατε σε σχέση με τις ε, εκκρεμότητες των πληρωμών και αυτά που μας εξηγήσετε πολύ λογικά μου φαίνονται. Ε, έχω να σας ρωτήσω το εξή. Ο πρόεδρος Ιούνκερ σας έστειλε μια επιστολή ανάθεσης καθηκόντων για την χάραξη προτεραιοτήτων στην αρχή για τις πληρωμές. Μπορείτε να μας δώσετε λίγες λεπτομέρειες, ποιες προτεραιότητες, πώς θα τις ορίσετε, με ποια κριτήρια και σε ποια βάση θα οριστούν όλα αυτά. Και δεύτερη ερώτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την αναθεώρησή του. Και ο κανονισμός λέει ότι οι εθνικές συνεισφορές για την συνοχή μάλλον κατανομή ένα κράτος, θα αναθεωρηθούν ε, ανάλογα με τις επενδύσεις, μάλλον στα κράτη δικαιούχους μετά το 2016. Για να υπάρξει ανάπτυξη φυσικά και θέσεις απασχόλησης σε αυτές τις χώρες. Στην πρώτη σας ερώτηση, έχω ήδη τονίσει οι ε, γενικές διευθύνσεις που δαπανούν χρήματα χρειάζονται μέτρα για να προγραμματίζουν καλύτερα και να εκτελούν τις πληρωμές. Στην ανθρωπιστική βοήθεια που είμαι αρμόδια ήμασταν οι πρώτοι που είδαμε αυτό το πρόβλημα, διότι στη δική μας περίπτωση αυξήθηκαν οι κρίσεις και αν δεν έχεις ε, να δώσεις λεφτό, ο κόσμος πεθαίνει. Οπότε ε, έπρεπε να συγκεντρώσουμε τις πιστώσεις πληρωμών και να τις διαχειριστούμε. Και τι κάνουμε, τα εξής τρία. Πρώτον, ε, προτεραιότητες είναι οι δραστηριότητες, οι δράσεις που σώζουν ζωές. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί να αναβληθεί και τι δεν μπορεί. δεύτερον, έχουμε διαρθρώσει τους εταίρους, τους έχουμε χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που ε, φέρουν μάλλον που μπορούν να αντέξουν μια πιο αργή ε, πληρωμή και εκείνους που επίγονται απολύτως. Ε, αν δείτε και στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών ε, στις προκαταβολές μας μειώσαμε το ποσό από 80% στο 40%. Μπορούν να το αντέξουν γιατί έχουν μεγάλη χρηματοδότηση. Για τις μικρότερες ΜΚΟ διατηρήσαμε το 80% για να μην αναγκάζονται να δανείζονται. Γιατί ε, πρέπει να επιβαρύνουν το φορολογούμενο και με την καταβολή ε, τόκων. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Να δούμε πώς εφαρμόζονται λοιπόν τα προγράμματα ε, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να δούμε πού μπορούν να υπάρξει αυτή η συνέργεια. Και το παράδειγμα, ας πούμε, στο Νότιο Σουδάν ε, ανέλαβε μεγαλύτερη οικονομική ευθύνη τώρα Άλλο εταίρου οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλού εμεί. Αυτό ε, είναι η φιλοσοφία μα γενικά. Βλαδιμίρ Μάνκα. Κυρία Γεωργίευα, αύξηση 16 στο 24 πήγε η ανεργία μεταξύ του 2007 και του 2013. Μιλάμε για πάνω από 15% αύξηση σε Ελλάδα και Ισπανία. Ποιος Γιούνκερ είπε ότι έχουμε μια ολόκληρη γενιά νέων οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν τη μάχη τους σε 29 κρατημένη. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε για αυτούς και για αυτούς που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Εσείς πώς εκτιμάτε το πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά ε, το, αυτό το πρόγραμμα ε, της εγγύησης για τους νέους. ότι το 2015 δεν θα υπάρχουν πλέον ε, πόροι για την του προγράμματος και εσείς τι προτείνετε ε, για την ιδέα να αυξηθούν ναι, τα χρήματα του προϋπολογισμού από το 2016 και μετά για να ε, πρικοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα για την νεολαία. Επίσης έχουμε κάποιους οργανισμούς που ζητούν για 21 δις για το 2014-2020 για αυτή την δουλειά, για αυτό το σκοπό. Εσείς τι λέτε όσον αφορά αυτό το ποσό. Σας ευχαριστώ κύριε Μάγκα. Αυτή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ήδη έχει αποδώσει καρπούς και μελετούσα για κάποιο είδου προγράμματα πάρα πολύ προχωρημένα σε κάποια κατημία Δεν ξέρω για την Ελλάδα, αλλά είδα ότι στην Γαλλία και στην Ισπανία είχαμε και στις δύο χώρες πάνω από 750.000 νέους οι οποίοι έχουν κάποια ευκαιρία να καταφέρουν κάτι ακριβώς λόγω του προγράμματος. Βεβαίω και εφόσον αποδίδει, εγώ 100% θέλω να υπάρξει παράταση και επέκταση. Να γίνει και αυτή η αναθεώρηση μεσοπρόθεσμη που είναι πολύ σημαντική. Γιατί Είπαμε να έχουμε κάποιο αποθεματικό όσον αφορά τι πιστώσει υποχρεώσεων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτέ τι πρωτοβουλίε, αλλά θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε περισσότερα για του νέου. Γιατί ε, είπα και το ξαναλέω, όντω όταν βλέπουμε τους νέους μας να μαζεύουν και να φεύγουν και να πηγαίνουν και να οδηγούν ε, άλλες χώρες πιο ανταγωνιστικές και προχωρημένες, αυτό είναι κάτι το θλιβερό. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Τώρα όσον αφορά τα 21 δις, πρέπει να το κοιτάξω και θα σας πω. Γιατί δεν έχω τόσο ξεκάθαρη εικόνα για το τι περιθώριο έχουμε και πόσο θα κοστίσει αυτή η προσπάθεια. Ακριβώς και αυτό θέλει να καταφέρει και ο κύριος Γιούγκερ. Θέλει να δώσουμε προτεραιότητα, θα αντιμετωπίσουμε αλλιώ, τι προτεραιότητέ μας όλοι μαζί, όχι ο κάθε επίτροπο χωριστά, όλοι μαζί θα ασχοληθούμε με αυτό. Γιάν... Ολμπριχτ. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας πω πρώτα απ' όλα ότι χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ μετά από πέντε χρόνια. Όντως, έχουμε καλή εμπειρία από εσάς και σας εύχομαι άλλα πέντε χρόνια επιτυχούς δράσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ήταν τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχετε λοιπόν μακρά εμπειρία και από τη συνεργασία σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μια πολιτική ερώτηση. Στις απαντήσεις σας μας είπατε τις απόψεις σας για την ε, μεταρρύθμιση των ε, διδαρτικών ταμείων. Θέλω να μας μιλήσετε για τις αλλαγές αυτές μέχρι το τέλος του 2016. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα και μεταξύ μας, γιατί θα υπάρξουν διαφορές. Γι' αυτό και είναι λίγο πρόκληση, προκλητική ερώτησή μου. Πάντως έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Πριν αναλάβετε τα καθήκοντά σας, από πού πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσετε και πότε. Απάντηση. Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν όλα πάνε έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί, 1η Νοεμβρίου θα αρχίσουμε και όχι αργότερα. Και ξέρω ότι είναι Σάββατο η 1η Νοεμβρίου. Δεν έχει σημασία. Γιατί δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε από την αρχή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την αναθεώρηση. Ξέρετε ότι δεν συμφωνούν όλοι με το στόχο. Κάποιοι λένε ότι ίσως να μην είναι καν πολιτικά εφικτό να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Μα θα γίνει εφικτή μόνο αν δουλέψουμε σκληρά για να έχει αξιοπιστία η πρότασή μας. Έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα από τις χώρες αυτές, οι οποίες ανησυχούν περισσότερο για το εγχείρημα, η άποψή τους είναι ότι έτσι θα δικαιολογήσουμε περισσότερες δαπάνες απλώς και μόνο και ότι δεν θα φροντίσουμε οι δαπάνες να γίνονται πιο ορθολογιστικά. Όμως η απάντηση που έχω να τους δώσω είναι το σχέδιό μας για απόδοση δαπανών. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να αποδεικνύει συνεχώς ότι οι δαπάνες μας είναι αποδοτικές και θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι σκεφτόμαστε το καλύτερο συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό από πίσω στους διαδρόμους. Το ξέρετε κι εσείς όμως, το ξέρω κι εγώ ότι θα είναι δύσκολο εγχείρημα. Αν όμως σκεφτούμε τι θέλουμε, ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε προτάσεις για επενδύσεις με 400 δισεκατομμύρια πιστεύω ότι θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Γιώργη Πυρίνσκι τώρα. Αξιότιμη κυρία Γεωργίευα, θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την εμπιστοσύνη με την οποία σας περιέβαλε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον προπολογισμό και τους ανθρωπίνους πόρους. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία και στην ακρόαση. Τώρα, στην Ένωση οι τεράστιες προκλήσεις που έχουμε είναι η αύξηση των ανισοτήτων και των αποκλήσεων τι θα κάνετε έτσι ώστε η πολιτική συνοχής να ασχοληθεί και να λύσει αυτό το πρόβλημα και να καταλάβουν οι χώρες ότι είναι προς όφελος όλων αυτό. Είναι μια τεράστια πρόκληση. Θα βοηθήσετε στις χώρες που υποφέρουν περισσότερο και που υπολείπονται να αυξηθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα. Και με τον Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο λογιστών να έχουν μια λιγότερο λογιστική και πιο ευρύτερη εικόνα της κατάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πυρίνσκι. Ε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα απαντήσω την ερώτησή σας στα βουλγαρικά με ιδιαίτερη χαρά και σας ευχαριστώ που έχω την ευκαιρία να το πράξω. Για να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν και οι διερμηνείς από τα βουλγαρικά. Έχω πάρα πολύ θετικές ε, προσδοκίες και ελπίδες να αποθέσει στην πολιτική συνοχής. Και η Επιτροπή σας θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία σε εκείνους που είναι σε λιγότερο καλή μοίρα να προχωρήσουν. Κάναμε προσπάθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι ε, 25% των πιο φτωχών περιφερειών απευθύνεται μέγα τμήμα των κονδυλίων της συνοχής. Και όταν ε, μιλούμε για τη μείωση του χάσματος και των ε, ανισοτήτων που δυστυχώς αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, δεν έχουμε υπόψη μας μόνο την πολιτική συνοχής αλλά και την πολιτική ανταγωνισμού. Και με το ε, έρασμο ΣΥΝ που είναι μέσα όλα αυτά που μπορούν να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες για νέους και επιχειρηματίες και νέους αγρότες. Χρειάζεται οπωσδήποτε οι νέοι μας να κυκλοφορούν ε, και να ε, προωθούν την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι διακαής μου πόθος στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να συγκεράσουμε αυτούς τους δύο στόχους. Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και χαμηλότερες ανισότητες και ε, αποκλήσεις. Έτσι είναι ένας πολύ παραγωγικός τρόπος πιστεύω να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάνιμπολ. Κυρία Επίτροπε. Όπως προείπατε, πολιτικές και προγράμματα θα πρέπει να αποδίδουν για όλους τους Ευρωπαίους και κυρίως αυτούς οι οποίοι παραδοσιακά είναι περιθωριοποιημένοι. Τι να κάνουμε σε κάθε επίπεδο, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μπορεί να κάνουν οι εθνικές αρχές, ούτω ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση των κοινωτικών πόρων, έχοντας υπόψη αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Και έτσι να έχουν προσθέμενη αξία και απόδοση και του τελευταίου ευρώ. Έχουμε την αναθεώρηση του καταστατικού για τους υπαλλήλους και έχει πολλούς στόχους αυτή η αναθεώρηση, αλλά βέβαια και καλύτερη απόδοση του προσωπικού. Εσείς πώς θα εφαρμόσετε αυτό το νέο καταστατικό, ούτως ώστε να αντιποχθήσετε τις προσδοκίες, ιδίως όσον αφορά τώρα την οικονομική συγκυρία, τη λιτότητα και των περικοπών έχουμε αυτή την πρωτοβουλία των 300 δις. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα έχουμε προσωπικό ποιοτικό και οι μειονότητε αλλά και οι γυναίκες θα ωφελούνται από την καινούργια διάρθρωση και θα έχουμε μακροπρόθεσμα αξιόλογα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Το νέο καταστατικό δεν είναι βάρος, σε διάφορους ε, τρόπους κατά τους οποίους το προσωπικό μπορεί να ποικίλει περισσότερο. Οπότε μέχρι σήμερα και Πρόκειται να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα αναπλήρωσης προσωπικού για λόγους ιστορικούς, διότι τα παλιότερα κρατημέλη έχουν συμβάλει και έχουν στείλει εδώ υπαλλήλους οι οποίοι τώρα συνταξιδοτούνται. Αλλά αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για το ίδιο το προσωπικό, του ίδιου υπαλλήλου, να γίνεται επομένω μια προσπάθεια προσλήψεων τέτοιων που να φέρνει περισσότερη ισορροπία αλλά και ποικιλία στο προσωπικό. Άρα έτσι θα πρέπει να συνεχίσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό αποτελεί και παράδειγμα για τα κράτη-μέλη. Αν εμείς έχουμε λοιπόν αυτή την πολυμορφία, την ποικιλία που θέλουμε, αυτό θα πρέπει να δικαιοτοπτρίζεται με τη σειρά του και στο τι κάνουν τα κράτη-μέλη για αυτές τις ενέργειες. Και έτσι να δούμε το πώς μπορεί να βοηθήσουν κάποια προγράμματα. Ένας τρόπος θα ήταν με το να στοχεύσουμε στους πιο περιθωριοποιημένους, σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, αλλά επίσης αποτελεσματικό είναι να καλύψουμε αυτές τις ε, ομάδες ε, στις πολιτικές μας το είπαμε και για ε, το να καλύψουμε τα δύο φύλλα. Οπότε έχουμε εκεί πρόγραμμα, στρατηγική που θα εφαρμοστεί, αλλά δεν είναι μόνο οι γυναίκες αυτοί που έχουν περιθωριοποιηθεί. Είναι, υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Δεν πρέπει να τους ξεχνούμε, θα αυτό θα ήταν ζημιά και απώλεια. Και για μας και για αυτούς. Άρα χρειάζεται αυτός ο μηχανισμός των αναφορών, εκθέσεων αλλά και των σεμιναρίων που ακολουθούν. Εδώ ολοκληρώνεται η σειρά ερετήσεων από την Επιτροπή Προπολογισμών και δίνω την Προεδρία στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Κύριε Σαβαρμά, πρώτος εξ του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Δικός μας ρόλος στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού είναι να διασφαλίζουμε ότι προστατεύονται καλά τα χρήματα των Ευρωπαίων. Πρέπει να πούμε στους πολίτες μας ότι χρησιμοποιήθηκαν σωστά τα χρήματά τους σε όλες τις χώρες μέλη. Και ξέρουμε ότι η εκτίμηση σφάλματος έχει αυξηθεί από το 2009 και ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές των χωρών μελών είχαν τη σωστή ενημέρωση από την αρχή. Παρ' αυτά ζήτησαν αποζημιώσεις. Σε 16% των συναλλαγών στην περιφερειακή πολιτική υπάρχει σφάλμα. Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα λοιπόν, πρέπει να υπάρξει το naming and shaming, να πούμε δηλαδή το ποιος φταίει και ας μην το ονομάζουμε έτσι το σύστημα, γιατί δεν υπάρχει ντροπή, να κατανομάζω και ντροπιάζω, δεν είναι θέμα ντροπή, αντίθετα. Συνεπώς κύριε Επίτροπε θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς είσαστε έτοιμοι να εντοπίσετε τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν και να τα αντιμετωπίσετε ώστε να απαλλαγούμε επιτέλους από αυτό το πρόβλημα. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, πολλές φορές σήμερα είπα ότι πιστεύω πως είναι ζωτική σημασία να λογοδοτούμε, να χρησιμοποιούμε σωστά τα χρήματα των φορολογούμενων και να το εξηγούμε αυτό κατανοητά και αποτελεσματικά. Το ποσοστό σφάλματος μου είπαν ότι φέτος αλλάζει η τάση και ότι θα υπάρξει μείωση. Να το δούμε. Το ποσοστό σφάλματος λοιπόν είναι πάνω από, 2% σε όλα τα κοινά προγράμματα. Από πλευρά της Επιτροπής, τα προγράμματα της Επιτροπής δηλαδή είναι κάτω από 2% εκεί το σφάλμα. Και χαίρομαι γι' αυτό. Πάντως, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην κοινή διαχείριση προγραμμάτων και κυρίως στις χώρες εκείνες όπου μένουν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Όχι απαραίτητα όταν είναι υψηλό το σφάλμα. Δεν δείχνει αυτό ότι δεν κάνουν καλή δουλειά οι χώρες. Μερικές φορές δείχνει ότι είναι πιο ειλικρινείς οι χώρες. Ότι κάνουν περισσότερες προσπάθειες στο να ελέγξουν και στο να μας ενημερώσουν για τα σφάλματα. Πάντως συμφωνώ μαζί σας ότι το να λέμε ποιος φταίει, να τον κατονομάζουμε, είναι κάτι που ήδη γίνεται και είναι σωστό. Αλλά όπως λέτε και εσείς δεν πρέπει να το λέμε κατανομάζω και ντροπιάζω. Το name and shaming τελικά μπορεί να στραφεί στο... σε ένα κρυφτούλι που θα παίζουν τελικά οι υπεύθυνοι και σε όλα μάλιστα τα επίπεδα. Συνεπώς η δικιά μου προσέγγιση είναι δώστε την πληροφορία, φροντίστε να προβληθεί μάλιστα, υπογραμμίστε την και δουλέψτε ώστε το μπορείτε πιο σκληρά ώστε να υπάρξει περισσότερη γνώση και περισσότερη κατανόηση του προβλήματος σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ Σοσιαλιστές και Δημοκράτες Κλέρ Μόντι. Ε, χαιρόμαστε ε, για τις απαντήσεις σας για την κρίση πληρωμών και ε, την δέσμευσή σας να παραμείνετε στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περασμένα χρόνια όμως οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο από τη μια το ε, Συμβούλιο και από την άλλη Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Από το προπολογισμό του 2011 οι συμφωνίες στη συνδιαλλαγή δεν μπορούν να θεωρηθούν ισόρροπες των δύο σκελών του προπολογισμού ε, η συμφωνία. Τις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αυτή η συμφωνία, τη δέχεστε, την απορρίπτετε. Δεν χωράει συζήτηση. Ε, υπάρχει πρόβλημα πληρωμών. Κάθε φορά ζητούν ε, τα κράτη διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Αυτό εμβαθύνει το ρήγμα δυσπιστίας και καχυποψία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα οι αρχαίοι κρατών και κυβερνήσεων παίρνουν κάποιες αποφάσεις, αλλά στη συνέχεια στη συνδιαλλαγή αυτά δεν μπορούν να ε, σταθούν. Ε, δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες μάχες. Χρειάζεται αλλαγή λοιπόν. Τι θα προτείνετε συγκεκριμένα για να έχουμε μια διαδικασία προϋπολογισμού πιο ομαλή και αποτελεσματική από την τόσο περίπλοκη όσο και ε, μακρά που έχουμε αυτόν τον καιρό. Αυτό το ερώτημα ελπίζω να μπορέσω να έρθω να σα το απαντήσω έχοντα ζήσει κάποιε από αυτέ τι διαδικασίε και τι διαπραγματεύσει και ήδη από αποκομίσω εμπειρία. Νομίζω ότι μπορούμε να εξορθολογήσουμε τη διαδικασία ε, κατάρτισης του προπολογισμού. Προς το παρόν, ειλικρινά, πρέπει ε, να μπω στις διαπραγματεύσεις, τα βαθιά, μέχρι τις 17-11 του πρέπει να έχουμε κάνει πρόταση και η διαπραγμάτευση γίνεται με διάφορες προτάσεις, με διάφορα νούμερα και ποσά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, αλλά το σημαντικότερο είναι το τελικό προφανώς. Τούν των λεχθέντων έχουμε ένα οξύτατο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε και συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για πιο ρεαλιστική και ορθολογική κατάρτιση του προϋπολογισμού. Εγώ προέρχομαι από μια μικρή γενική διεύθυνση που δαπανά χρήματα από τον προϋπολογισμό και είναι πραγματικά πολύ περίπλοκο αυτό το εγχείρημα και όχι απαραίτητο αυτό που θα κάναμε εμείς αν ακολουθούσαμε καλύτερη διαχείριση ή χάραξη στον προπολογισμό. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, υπάρχει το ιστορικό, πώς θα βγούμε από αυτό. Ε, αυτό είναι το ζήτημα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω το πιο εύκολο σκέλος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα. Και αν ε, έρθουμε με ένα κοινό στόχο, και πούμε μια στιγμή, ας επικρατήσει λίγο η λογική εδώ πέρα. Ας δείξουμε καλή θέληση. Πάλι πέρασα το χρόνο. Τελειώνω λέγοντας ότι δεν το βάζω ποτέ κάτω. Ε, ECR Anders Vistisen. Κύριε το ECR ε, σέβεται τα χρήματα των φορολογουμένων τα οποία εμείς εδώ διασπαθίζουμε ή ξοδεύουμε απλώς. Οπότε πέστε μας, θα μπορέσετε να ε, ξοδεύσετε τα χρήματα με σοβαρότητα. Είχαμε το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο κάθε χρόνο επισημαίνει το πώς διασπαθούνται τα χρήματα και δεν έχουν προστιθέμενη αξία για αυτές ε, τις δαπάνες. Και θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των διασυνοριακών έργων υποδομής και αυτών που επισημαίνει το ελληνικό συνέδριο ως ε, αχρίαστες δαπάνες. Μπορείτε εσείς να κάνετε περικοπές, πού θα τις κάνετε, θα τις κάνετε σε όλες τις πολιτικές ή εκεί που δεν ε, πιάνουν τόπο οι τα χρήματα που ξοδεύουμε θα πάνε. Επιτροπος, δεν ξέρω αν κατάλαβα όλα όσα είπατε. Με ρωτάτε το πως θα κάνω περικοπές στον προϋπολογισμό σας απαντώ ότι ο προϋπολογισμός είναι προϊόν διαπραγματεύσεων. Και η δουλειά μου είναι να τον εκτελέσω και τον εκτελούμε όσο καλύτερα μπορούμε τον προπολογισμό. Αλλά βεβαίω θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί σε αυτή τη διαχείριση για τι τεθήσει προτεραιότητε μήπως τυχόν και δεν πιάνουν τόπο. Οπότε θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κατάλληλες αλλαγές. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Ακριβώς για τα όσα είπαμε για την προηγούμενη ερώτηση, για το ότι η διοργία του προβολισμού είναι πάρα πολύ περίπλοκη και έχουμε ένα σωρό παραμέτρους στις ε, υποχρεώσεις μας, οπότε θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει μια δύσκολη ενδελεχής διαχείριση του προπολογισμού. Πάντως συνεργάζομαι με το Ελληνικό Συνέδριο πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις συστάσεις και ελέγχους που κάνει το Ελληνικό Συνέδριο και το Συνέδριο επίσης ε, ενδιαφέρεται για να είναι αποδοτικές, αποδοτική η έλεγχη που ασκεί. Ξέρουμε επίσης τι γίνεται με το επίπεδο για το ποσοστό των λαθών. Αυτό τι είναι. Είναι ένα ποσοστό. Ποσοστό που αφορά, όπως λέει η ετύπωση, τα λάθη. Από το 4,8 μόνο το 0,2 ευτυχώς αφορούσε απάτες για πέρσι αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, το 0,2% και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αφόρετο και απαράδεκτο. Όμως, πολλές φορές θα πρέπει να προσέχουμε πώς ερμηνεύουμε κάποια στοιχεία. Πάντως, εμείς αυτό έχουμε ως ε, μέσο μέτρηση κατάστασης και πρέπει να βελτιώσουμε τη μέτρηση της κατάστασης. Κύριε Υποψήφια Πίτροπε, στην γραπτή σας απάντηση λέτε ότι θέλετε να εξηγήσετε καλύτερα την πραγματική αξία του ευρωπαϊκού προπολογισμού και να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τον προπολογισμό για τις ψηφιακές τεχνολογίες, λέει η κυρία Κάλλας. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξή. Ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβετε τον πρώτο χρόνο της εντολής σας για να πετύχετε αυτό το στόχο. Και δεύτερον, τι μέτρα θα πάρετε για να βελτιώσετε παρετέρω την πρόσβαση στα μέτρα αυτά για βελτίωση της απόδοσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Απάντηση. Τον πρώτο χρόνο θα αρχίσω από τις γενικές διευθύνσεις, οι οποίες αναφέρονται απευθεία σε μένα. Και θα δω τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να βελτιωθεί το σύστημα διαφάνειας και ενημέρωσης προς το κοινό. Πολλά μπορούν να γίνουν για να έχουμε διασύνδεση των βάσεων δεδομένων που ήδη υπάρχουν και πολλά μπορούν να γίνουν για να απλοποιήσουμε την ενημέρωση προς τα έξω. Η τεχνολογία λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά η τεχνολογία δεν πρόκειται να λύσει τα θέματα τα ενιολογικά. Τεχνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι υψηλών προσόντων και δίνουν την ενημέρωση στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι με αντίστοιχα προσόντα. Οπότε χρειάζεται κάποια ερμηνεία. Όχι η γλωσσική, έτσι, όχι η ερμηνεία, ενώ τεχνικά πρέπει να απλοποιηθεί η γλώσσα. Αυτή τη βελτίωση πρέπει να δούμε πώς θα την κάνουμε, να την κοστολογήσουμε πρώτα απ' Σκοπεύω πάντως να προσπαθήσω να βρω τρόπους όπου η πρόσβαση στην ενημέρωση από το κοινό να βελτιώνεται. Και δεν θα βελτιωθεί μια και έξω, εν μια ανοιχτή. Είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή την πληροφορία πιο αποτελεσματικά, ώστε να φτάνει πραγματικά στο κοινό και το κοινό να καταλαβαίνει τι κάνουμε και να έχει νόημα το ότι λογοδοτούμε. Πριν από λίγο καιρό έψαχνα κάτι στο διαδίκτυο και στο τέλος σήκωσα τα χέρια ψηλά. Μα δεν γίνεται. Τον πρώτο χρόνο λοιπόν θα επικεντρωθώ στη δικιά μου την ομάδα, τι κάνουμε εμείς και μετά θα προσπαθήσω αυτό να το επεκτείνω και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Ευχαριστούμε. Διάφορες επιχειρήσεις παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μετεγκατασταθούν. Είναι παράδεκτο, όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι πολίτες να πληρώνουν γι' αυτό και το έχει πει αυτό και ο προκάτοχός σας. Και το πρόβλημα το διαπιστώσαμε όταν κοιτάξαμε τι γίνεται με τις καταχρήσεις και είδαμε ότι είναι μια ε, παραβίαση που γίνεται και το διαπιστώσαμε όταν αναγκάστηκαν να κάνουν δηλώσεις όσες επιχειρήσεις είχαν πάρει χρήματα από τον κοινοτικό κορβανά. Τι θα κάνετε λοιπόν ώστε να μην πηγαίνουν ευρωπαϊκά χρήματα σε επιχειρήσεις οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρονται από μια ευρωπαϊκή χώρα ε, αλλού. Έχετε, σκοπεύετε να φτιάξετε έναν, μια μαύρη λίστα με τέτοιου είδους επιχειρήσεις που μετακαθίστανται. Ευχαριστώ. Απάντηση. Δεν ε, είμαι εξοικειωμένη με το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναφέρατε, θα το κοιτάξω για να μπορέσω να σας απαντήσω πιο συγκεκριμένα. Γενικά μιλώντας πάντως, άπαξ και κάποιος παίρνει χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και δεν τα χρησιμοποιεί σωστά, αυτό πρέπει να διορθώνεται για να το πω με απλά λόγια. Αν παίρνετε χρήματα για να τα χρησιμοποιήσετε για ένα σκοπό, πρέπει να πηγαίνουν σε αυτό το σκοπό. Άρα πρέπει να γίνουν διορθώσεις, οι οποίες μάλιστα ε, λειτουργούν και αποτρεπτικά ώστε να μην το κάνουν κι άλλοι. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω το συγκεκριμένο θέμα. Θα φροντίσω εδώ οι συνεργάτες μου να το σημειώσουν και θα επανέλθω σε εσά απευθείας αργότερα. Ο Μπάρτης Στάς από τους Πασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ε, εκφράσω την εκτίμησή μου και την αναγνώριση όπως όλοι για το έργο σας την τελευταία πενταετία και είμαστε σίγουροι ότι θα αφοσιωθείτε πλήρως στα νέα καθήκοντα. Στην ε, γραπτή σας απάντηση και δήλωση λέτε ότι θέλετε μια όλα αυτό ε, κατά της απάτης που να είναι αυστηρή, αποτελεσματική και να γίνεται και σεβαστή. Συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Πρώτον, τα αποτελέσματα του Όλαφ δεν είναι μπορούν να εξακριβωθούν ή να επικυρωθούν με σωστό τρόπο και γίνεται και μια συμφωνία, συζήτηση μάλλον με τον τρόπο που δίνει τα στοιχεία. 99% του προσωπικού της Όλαφ ψάχνει άλλη δουλειά. Δηλαδή δεν τους αρέσει εκεί που δουλεύουν. Και υπάρχει και μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στην Εποπτική Επιτροπή, το Εποπτικό Συμβούλιο και την Όλαφ την ίδια. Και ο σημερινός διευθυντής δεν επιτρέπει ε, ε, ισχυρούς ελέγχους και αποτελεσματικούς. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Απάντηση. Για μένα ε, όλο αυτό το γραφείο κατά πολέμησης απάτης δεν είναι σημαντικό μόνο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που είναι η βασική του αποστολή αλλά και από πλευρά πολιτικής διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο απέναντι στα κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζετε, η θητεία μου και η εντολή μου για την Όλαφ είναι ξεκάθαρη και πολύ καλά ορισμένη. Έχω ευθύνη ε, όχι όμως για την πλευρά της έρευνας η ανεξαρτησία ε, τη Όλαφ είναι εκ των όνων κάνευ. Και εγώ θα ήμουν η τελευταία που θα έκανα το παραμικρό που με οποιοδήποτε τρόπο θα ε, έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να ε, υπερβαίνω τα εσκαμμένα της δικής μου εντολής και ευθύνη. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ ως αρμόδια για τις πολιτικές είναι να συνεργαστώ πολύ στενά με την Όλαφ και να δω εάν έχουμε τις σωστές προτεραιότητες, τι κάνει από πλευράς πολιτικής, πώς μπορεί να βελτιωθεί και η στρατηγική κατά των ε, προβλημάτων διαφθοράς στα κράτη-μέλη κτλ. Και δεύτερον, ε, αν επιβεβαιωθώ ως αντιπρόεδρος αρμόδια για τους ανθρώπινους πόρους, ανησυχώ ε, από τα αποτελέσματα της έρευνας στην Όλοφ, αλλά αυτό ισχύει και για άλλες γενικές διευθύνσεις και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να παρακολουθήσω και να δώσω συνέχεια τι μέτρα ελήφθησαν εκεί, τι μέτρα ελήφθησαν αλλού. Θα είμαι πολύ προσεκτική. Γιατί πραγματικά εγώ θέλω το προσωπικό μας να μπορεί να ασκεί τα υψηλά καθήκοντα που του ανατίθενται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε ένα ε, περιβάλλον ε, ωραίο και στο οποίο αισθάνονται άνετα για να εργάζονται. Ο Μάρκο Βαλέ από το EFTD. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Διάβασα τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που σας υπέβαλε το Κοινοβουλίο και μου αρέσει το ότι θέλετε να καταπολεμήσετε διαφθορά και απάτη γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το θεμέλιο για κάθε όργανο το οποίο διαχείριζεται δημόσιο χρήμα θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση και διαφάνεια. Ξέρετε, στην Ιταλία έχουμε το πρόβλημα της Μαφία και έχουμε ένα σωρό έρευνες και ανακρίσεις από τις αγγελικές αρχές είναι ένα πρόβλημα διαρθρωτικό για μας και είναι πρόβλημα αυτό για τον Ιταλό φορολογούμενο γιατί έχουμε μία από τις πιο ψηλές φορολογίες στον κόσμο και πληρώνουμε την ύφη τελικά εμείς για αυτό τόσο, το τόσο βαθύ φαινόμενο της ε, μαφίας και της διαφθοράς. Εσείς θέλετε να δεσμευτείτε για το ότι θα βοηθήσει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχουν λαθροχειρίες ε, σε σχέση με τις μαφίες στα κρατημέλη. Βεβαίως, κατηγορηματικά σας το καταφατικά. Διότι παρακολουθούμε στενά το πώς ε, γίνεται η διαχείριση των πόρων μας και προσπαθούμε πριν παροξενθεί το πρόβλημα να κάνουμε κάτι. Πέρσι η Όλαφ μετά από έρευνε ανέκτησε 117 εκατομμύρια ευρώ που είναι πολύ σημαντικό ποσό όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτό σας δείχνει το πόσο σοβαρά βλέπουμε το πρόβλημα της ανάκτησης ε, των ε, πόρων. Βέβαια δεν πρόκειται πάντοτε για διαφθορά, για κλιματική ενέργεια, απλώ πολλές φορές είναι λάθος, είναι τέλος πάντων παρατυπία, κάποιος δηλαδή παίρνει τα χρήματα γιατί αν τα πάει για αυτό στο οποίο προορίζεται, τα κάνει κάτι άλλο, αλλά το άλλο αυτό είναι κάτι το θεμητό. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Βέβαια με το φαινόμενο αυτό στις χώρες, αλλά και οι ίδιες χώρες θα πρέπει να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Ίσως όλοι εδώ έχουμε δει έργα, πολλά έργα στον κινηματογράφο για την μαφία. Από την άλλη μεριά όμως δίνουν σκληρή μάχη οι δικαστές, οι εισαγγελίες, έτσι κάνοντας τη ζωή τους στη χώρα σας. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, τους υποστηρίξουμε. Είναι υποχρέωσή μας αυτή. Να, είδατε καμιά φορά σταματάω και πριν λήξει ο χρόνος. Είδατε. Και έτσι τις περιβάσεις τις ξεπληρώνω τώρα. Λουί Αλιό, Λουί μη Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλήσατε προηγουμένως για τα αποτελέσματα που ε, πετύχατε. Ναι, αλλά κοιτάξτε σε σχέση με τα ευρώ που δίνουμε και τα πόσα ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι οι πολίτες των κρατών μελών μας χάνουν την εμπιστοσύνη σου στην Ευρώπη. Όλοι Ευρωπαίοι είμαστε, αλλά σε αυτό το σύστημα δεν εμπιστεύονται πια το σύστημα οι Ευρωπαίοι. Και σε αυτή την ε, απώλεια της εμπιστοσύνης πιστεύω ότι είναι πλήρης η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δώσατε ένα παράδειγμα συμπαθητικό για το μετρό της πόλης που ζείτε, ότι τη χρηματοδοτεί η Ευρώπη. Να σας πω, εγώ από εκεί που έρχομαι, η ευρωπαϊκή πολιτική κάνει μεγάλες ζημίες με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων που επιτρέπει στο εσωτερικό της Ένωσης στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ε, που ε, κάνουν ανέργους τους εργαζόμενους και τις εταιρείες να πτωχεύουν. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα σήμερα από όσα λύνει και μπορεί κάποιους να καθιστά ευτυχής αλλά κάποιους άλλους κάνει δυστυχέστατος. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπω να προβληματίζεστε, στη συνείδησή σας δηλαδή κατά πόσο λειτουργεί σωστά η Ένωση. Και θέλω να σας ρωτήσω για την απάτη, τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή με συγκεκριμένο παράδειγμα. Πρώτον, η κακή πληροφόρηση όλα το χρόνο σας. Δεν κάνω την ερώτησή μου, Πρόεδρε. Το σκάνδαλο, για παράδειγμα, στην Καταλωνία, όπου ένας ε, Ισπανός πολιτικός ε, πήρε χρήματα από την Ευρώπη και τα πήγε στην Ανδόρα. Τι σκέφτεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Obviously, Προφανώς πάντα στόχος είναι να βελτιωνόμαστε και στις πολιτικές μας και στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογμένων. Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχουν ορισμένοι στην Ευρώπη που θεωρούν ότι ορισμένες πολιτικές, ιδιαίτερα η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ε, προκαλεί προβλήματα τοπικά. Αλλά θα πρέπει να δούμε και τα ωφέλη από την ελεύθερη κυκλοφορία προς τα κράτη-μέλη. Και τα ωφέλη είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Πέρα από όλα αυτά όμως, και το ειδικό πρόβλημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Θα πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να βλέπουμε τι γίνεται και στον έξω κόσμο και να αναγνωρίσουμε ότι από την σκοπιά της ανταγωνιστικότητας είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε για να έχουμε μια οικονομία που είναι αρκετά μεγάλη ως οικονομία κλίμακος και ως αγορά για να μπορούμε να είμαστε ακόμα ανταγωνιστικοί. Είμαστε ακόμα υπαριθμόν ένα οικονομία παγκοσμίω, πάνω από 20% του ΑΕΠ. Είναι δικό μας, του παγκοσμίου. Το μερίδιο μας όμως συρρυκνώνεται και ο κόσμος δεν πρόκειται να ζει καλύτερα αν δεν αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Με χώρες μικρές που να ακολουθεί κάθε μια το δρόμο της. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τρόπος να βελτιωθεί η ζωή μας. Το συγκεκριμένο παράδειγμα που μας αναφέρατε δεν το γνωρίζω. Θα ενημερωθώ και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα ερχόμαστε στους ομιλητές ε, των πολιτικών ομάδων, το Μαστόιτσο από το ΕΛΚ. Η τελευταία έκθεση απαλλαγή ζητάει δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ε, λυθούν οι επιφυλάξεις της τελευταίας έκθεσης κυρίως για τα διευθυντικά ταμεία. Διάβασα τις απαντήσεις σας, τις γραπτές, αλλά αναρωτιέμαι ακόμα πώς μπορεί κανείς πιο γρήγορα και πιο εύκολα να αντιμετωπίσει τα θέματα παρατυπιών. Να έχουμε μηδέν ανοχή. Επίσης, η ερώτησή μου έχει ως εξής. Τι θα κάνετε προκειμένου να επικεντρωθείτε στα πραγματικά προβλήματα που βρίσκουμε μπροστά μας, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντιμετώπισης των ατασταλιών και των παρατυπιών. Να λυθεί ο χρόνος δηλαδή επεξεργασία τους και αντιμετώπισης τους. Θα παγώσετε πληρωμός, πληρωμές εφόσον επανειλημμένα ε, παρατηρούνται καταχρήσεις ή παρατυπίες από τους ίδιους. Απάντηση. Μηδέν ανοχή στην απάτη. Μηδέν, μηδέν, μηδέν. Και πάλι, αν υπήρχε και χαμηλότερο νούμερο από το 0, θα το αυτό. Είναι πραγματικά δηλητήριο, καταστροφικό το να ανέχεται κανείς απάτες. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τις δύο ερωτήσεις σας, έχω να σας πω το εξής πηγαίνουμε σε ένα σύστημα ελέγχου που να βασίζεται όλο και περισσότερο στις πιθανότητες κινδύνου και στην επανάληψη κινδύνου. Και προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίε τους και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε τη βοήθεια του ελεκτικού συνεδρίου, του δικού μας εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των γενικών διευθύνσεων που κάνουν τις δαπάνες. Πρέπει να απλοποιήσουμε πάντως τους κανόνες γιατί όσο πιο απλοποιημένοι είναι τόσο πιο πολύ θα συμμορφώνονται οι άνθρωποι. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ στην Κομισιόν όσο στις χώρες μέλη που εφαρμόζουν όπως εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μερικές φορές αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο είχαμε περισσότερα σφάλματα. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για το πάγωμα, βεβαίως, ιδιαίτερο όταν πρόκειται για επανάληψη παρατυπιών ε, και απατών. Κυρίως όταν θα μπορούσαν να το έχουν προβλέψει ή το ξέρανε και δεν κάνανε τίποτα. Τότε ναι. Διότι από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Δώσατε τι απαντήσει στο ερωτηματολόγιο και εκεί αναφέρατε ότι για σας είναι κορυφαία προτεραιότητα το τι θα κάνετε με την κρίση όσον αφορά τι πιστώσει των πληρωμών. Είπατε ότι θα λάβετε υπόψη το προσχέδιο προπολογισμού 14-15. Ε, ε, σας ερωτώ, η Ευρωπαϊκή μπορεί να μας εγγυηθεί εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο ότι πρόκειται να μείνετε πιστοί ε, σε αυτά τα οποία είπατε στη συνδιαλλαγή, ε, αυτά τα οποία τότε προτείνατε προς εμάς. Άλλη ερώτηση. Τα κράτη-μέλη υποτιμούν όλο ένα και περισσότερο το ότι ο προϋπολογισμός είναι ε, όργανο διακυβέρνησης, οπότε όλο ένα και περισσότερο μειώνουν τους πόρους για την ανάπτυξη. Ε, εμείς εδώ πολλές φορές έχουμε πει ότι θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή την τάση όταν αξιολογεί το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τι εισφέρουν τα κράτη-μέλη. Εσείς τι προτείνετε ούτως ώστε να μπορέσουμε να μπορέσετε να καλύψετε το αίτημά μας. Επίσης, πώς θα συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας, κυρίως με τον κύριο Ντομβρόφσκι και τον κύριο Μοσκοβεσί για τα θέματα επί των οποίων σας επέβαλα ερώτηση. Γεωργίευα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να διευκρινίσουμε όταν ε, είπατε κυβέρνηση εννοείται εθνική κυβέρνηση ή τοπικές αρχές. Α, εθνικές ε, κυβερνήσεις. Τα εθνικά κοινοβούλια για να αρχίσουμε από το προφανές όντως υποβάλλουν αυτές τις δηλώσεις αξιοπιστίας. Και εμεί θέλουμε σε αυτήν την υπόθεση να εμπλέξουμε εθνικά κοινοβούλια. Τώρα, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα προγράμματα που ε, εμείς προτείνουμε και τρέχουμε. Εκεί όντω έχουν προταθεί κάποιες περικοπές, ιδίως όσον αφορά κάποιες διοργανικές σχέσει που δεν αφορούν μόνο τα θεσμικά όργανα, αφορούν και τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών. Οπότε και η Επιτροπή έχει αυτό το τιτάνιο έργο του να μπορέσει να εμπλέξει πιο άμεσα τα θεσμικά όργανα. Γιατί εδώ τα βρίσκουμε, τα συμφωνούμε, αλλά ο κόσμος είναι στα κράτη-μέλη. Ο κ. Σπυρίνσκι ήταν συνάδελφος στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο και ξέρει τι έγινε εκεί, πώς ενεπλάκει δηλαδή το Εθνικό Κοινοβούλιο επανειλημμένα και πόσο σημαντικό είναι βέβαια κάτι τέτοιο. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά τα προγράμματα και τις τοπικές αρχές. Έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις και είπατε σωστά ότι δεν ξέρετε αν εμείς θα εμείνουμε στην πρότασή μας. Βεβαίως και θα είμαστε σταθεροί σε αυτό το οποίο προτείναμε. Η Επιτροπή υπευλώθηκε την πρόταση, όχι τυχαία, αλλά κατόπιν πολύ σοβαρής αξιολόγησης. Γιατί ήταν σημαντικά τα προβλήματα και σημαντική η κίνδυνη και όλα αυτά τα παρακάμψαμε. Τέλος πάντων, μην τα ξαναπούμε, γιατί τέλειωσε ο χρόνος. Ο Γιάννη Κερπράντη, ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να τονίσω ότι προσβλέπω πάρα πολύ στη συνεργασία μαζί σας τα επόμενα έτη στο προπολογισμό και τον έλεγχο προπολογισμού. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή δηλώνεται ε, ότι θέλετε να ε, αλλάξτε την εστίαση προς τα αποτελέσματα. Χρειάζεται οπωσδήποτε. Το ελεγκτικό συνέδριο το έχει πει επανειλημμένα και πάρα πολύ στεναρά και παγίως τα αγνοούν τα κρατη και πολύ συχνά δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα παράδειγμα, 5 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για τη βιομηχανία τροφίμων, μία ενίσχυση που δεν ε, ε, είχε προστιθέμενη αξία, γνώρισε σφοδρή κριτική και έπρεπε να είχε σταματήσει. Τι θα κάνετε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα πιέσετε τα κράτη-μέλη να εστιάζουν πολύ περισσότερο στην αποτελεσματικότητα γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ επίσης και για την ε, προσφορά για περισσότερη συνεργασία ε, και εγώ προσβλέπω πάρα πολύ σε αυτήν. Πραγματικά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κοιτάξετε το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ουσιαστικά αυτό που την ενδιέφερε ήταν η νομοθετική εναρμόνιση. Αποτέλεσμα. Έχουμε εξαιρετικούς δικηγόρους, κατά κύριο λόγο. Αυτό μας που χρειαζόμαστε τώρα είναι ανθρώπους που να έχουν πιο οικονομική σκέψη και ε, περισσότερο δημοσιονομική. Τους ε, προσλαμβάνουμε τώρα. Όταν είσαι δικηγόρος, ε, σε ενδιαφέρει πιο πολύ η διαδικασία, ενώ όταν είσαι οικονομολόγος, ας πούμε, σε πάρα πολύ περισσότερο για το αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα ολόκληρη και παρακαλώ μην με παρανοείστε. Ε, και βεβαίως χρειαζόμαστε δικηγόρους και δεν θέλω να τους καταργήσουμε γιατί είναι και η καθημερινή μας ζωή αυτή. Αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να επιταχύνουμε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας και εστίασης. Και αυτό θα γίνει μόνο αν όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συνεχίσει αυτό με συνέπεια. Ε, με ρωτήσατε τι θα κάνουμε. Δεν είχα χρόνο να απαντήσω. συγγνώμη. Συνεργασία με τους επιτρόπους που ασχολούνται με χαρτοφυλάκια που έχουν δαπάνες για να μετρήσουμε και την πρόοδο που θα γίνει εκεί και να τη μετρούμε συχνά σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Κύριε Επίτροπε, από το ΕΛΚ θα μιλήσω εγώ και θα κάνω και εγώ μια ερώτηση. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της Όλαφ που έχει προβλήματα στη λειτουργία. Τα δύο τελευταία χρόνια το Εποπτικό Συμβούλιο κατέδειξε προβλήματα και παρατυπίες και ατασταλίες ε, κατάχρηση εξουσίας, παράνομες ε, έρευνες, ε, υπάρχει και ποινική συνέχεια. Τα αποτελέσματα αυτά της εργασίας είναι και το γεγονός γιατί δυσκολεύουν τώρα τη ζωή του Επιπτικού Συμβουλίου. Ο νυν επίτροπος για την καταπολέμηση της απάτης δεν ενδιαφερόταν πάρα πολύ και ε, οι δικές απαντήσεις ήταν κάπως ασαφείς. Εσείς θα συνεχίσετε τον δρόμο που χάραξε εκείνο και θα είστε έτσι απλή παρατηρήτρια ή θα κάνετε τίποτα διαφορετικό τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Uh, the... Απάντηση. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου για την ακρόαση, όχι μόνο από τις ερωτήσεις και από άλλες ε, συνεδριάσεις κατάλαβα ότι υπάρχει αυτή η ένταση μεταξύ Όλαφ και Εποπτικής Επιτροπής. Δεν είναι κακό να υπάρχουν εντάσεις, μπορεί να είναι και δημιουργική ένταση, μπορεί να διαπληκτίζεσαι, να διαφωνείς και να υπάρχουν εγώνιμες στη συνέχεια αλλαγές. Σήμερα δεν είμαι σε θέση να κρίνω τι τρέχει. και δεσμεύομαι πάρα πολύ από τους περιορισμούς του δικού μου ρόλου. Γιατί η Εποπτική Επιτροπή και Όλαφ έχουν το ερευνητικό σκέλος όπου εγώ δεν έχω κανένα ρόλο. Εγώ κοίταξα τα θέματα που έχω λόγο και ρόλο, ας πούμε τη στελέχωση. Η Εποπτική Επιτροπή έχει ενισχυθεί σε ανθρωπίνους πόρους για να υποστηριχθεί. Και επίσης ξέρω ότι υπάρχει και ένα θέμα ε, για το που βρίσκεται ο προϋπολογισμός και το προσωπικό τους. Αυτό είναι περισσότερο στα δικά μου χωράφια. Αλλά αν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός. Αξίζει τον κόπο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα συνεχίσω πολύ προσεκτικά να αξιολογώ τα πράγματα που εμπίπτουν στη δική μου αρμοδιότητα. Και πάλι με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί αν δεν διαφυλάξω εγώ την ανεξαρτησία του όλα, ποιος θα το κάνει. Στα πλαίσια λοιπόν των αρμοδιοτήτων μου και των ευθυνών μου θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι όλα αυτά διατηρήσει την ε, φήμη που έχει, το ρόλο που έχει και το έργο που κάνει που είναι τόσο σημαντικό για όλους μας. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η κυρία Γιάλα Σέντερ. Eh, Ευχαριστώ, κυρία Γιώργεβα. Αναφερθήκατε στο θέαμα το διακυβερνητικό που κάθε 7 χρόνια όλο και λιγότερο κοινοτικό προπολογισμό εγκρίνουν όπως έγινε και την τελευταία φορά και που λιγότερο προστατεύει τελικά τους ε, πόρους. Πρέπει όμως να ξεφύγουμε από τους εθνικούς εγωισμούς. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να πετύχουμε πραγματικά κοινοτικού ιδίω πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που βρίσκονται σε κρίση. Ακούσαμε αυτά που μας είπατε, ακούσαμε και τον κύριο Γιούνκερ για το βάρος των οικονομικών μέσων που πρέπει να αυξηθεί βάσει διαφόρων πολλαπλασιαστών και έτσι έχουμε καταλήξει σε μια, πώς το τραπεζική διάσταση ας πούμε του κοινοτικού προϋπολογισμού. Εντάξει, το λέω κάπως αστεία, αλλά δεν θα ήθελα να γίνουμε τράπεζα και εμείς στο μέλλον. Στην πραγματική οικονομία όμως, όλα αυτά τι αντίκτυπο θα έχουν. Έπειτα, λέτε ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην ομάδα προβληματισμού για τους ιδίους πόρους. Και εμείς πρέπει όντως να υπάρξει νέα ε, διάσταση στους ίδιους πόρους. Τι θα κάνετε επίσης για να καλύψετε τις απώλειες που από ό,τι φαίνεται απορρέουν από τα τελωνία μας όπως ε, έχει ακουστεί τελευταία. Ευχαριστώ. Απάντηση. Για το πρώτο, για τους ίδιους πόρους. Είναι τυχές, πραγματικά. Με έθλιψε πολύ το γεγονός ότι κατέληξαν διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι όπως κατέληξαν. Θα έπρεπε να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό καλύτερα αντικυκλικά από ό,τι κάναμε τώρα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, το κάναμε, αλλά η απόφαση είναι αυτή που είναι. Πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στο να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν θέλω καθόλου να κάνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τράπεζα. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο κάτω-κάτω. Θα ήθελα όμως να δω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί τους οικονομικούς της πόρους με περισσότερη φαντασία. Γιατί και το δεχόμαστε όλοι αυτό, ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να καλύψουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες. Και αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα με τα χρήματα που έχουμε, τότε πρέπει. Αν δείτε τους στόχους για τα διάφορα προγράμματα, αν σκεφτούμε με περισσότερη φαντασία, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με τέτοια χρήματα. Γιατί με την φαντασία μας θα βρούμε περισσότερους τρόπους και διαφορετικούς τρόπους ώστε να αποδώσουν περισσότερο οι προσπάθειές μας. Όσον αφορά τώρα τους ίδιους πόρους. Ναι, το λέω και το ξαναλέω ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα ιδίων πόρων. Αλλά τελικά είναι πολιτική επιλογή. Συνεπώς πρέπει να πιστούν όσο γίνεται περισσότεροι. Μερικές φορές στην Ευρώπη δεν τα καταφέρνουμε. Αλλά θα το κάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Ολοκληρώνεται εδώ και ακολουθεί η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Α, ξέχασα την κυρία Σμίτ όμω που ήταν ακόμα τη Επιτροπή Ελέγχου, λέει η Πρόεδρος. Βιάζομαι. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν το 2011 ε, ε, έκρινε ένα πακέτο για το προσωπικό ένα δισεκατομμύριο μέχρι το 2020 μπορεί να ε, εξοικονομήσει και μετά ένα δισετησίως. Και μέχρι το 2020 παγώνουν οι διοικητικές δαπάνες. Οι συνολικές δαπάνες είναι 5,8% του συνολικού προϋπολογισμού. Εξών 40% για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η συμφωνία σημαίνει ότι μέχρι το 2020 κατά 5% πρέπει να μειωθεί το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερωτώ πώς θα υλοποιήσετε αυτό το στόχο, με ποια συγκεκριμένα μέτρα, πώς έχει το χρονοδιάγραμμά σας και πώς θα μετρηθεί η επιτυχία των μέτρων. Και θα μας ενημερώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ. Uh, it is, uh, thank you. It is... Σας ευχαριστώ κύριε Γεωργίευα. Βέβαια, βέβαια. Ακριβώ η αξιοπιστία μα έγκυται επιτοπλίστων σε αυτό το να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχόμαστε και αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία έτσι θα πρέπει να κάνουμε και αυτό το 5% ε, ε, περικοπή είναι κάτι το οποίο ε, θα το κάνουμε γιατί τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια ανακατονομή των θέσεων ούτως ώστε να υποστηρίξουμε κάποιες υπηρεσίες που έχουν υψηλή προτεραιότητα εις βάρος κάποιων που δεν έχουν υψηλή προτεραιότητα. Ας πούμε τα χρηματοοικονομικά έχουν 30% αύξηση σε προσωπικό παρά τη γενικότερη περικοπή. Οπότε για να σας απαντήσω όσον αφορά τις προσλήψεις και λοιπά έχουμε ε, όλοι μαζί ενεργούμε, τα συζητάμε, με τι χρήματα υπάρχουν γιατί αν γίνει αναλογικού είδους ε, περικοπή ε, δηλαδή αν κόψουμε τα ίδια από παντού, ε, τότε αυτό θα δυναμητήσει το έργο μας, δεν το θέλουμε. Και επίσης θα πρέπει να δούμε, να, να, να, έχουμε, να κάνουμε προγνωστικά, τι, τι, τι θα βρούμε μπροστά μας κατά κάποιο τρόπο. Ε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένε δεξιότητες, γιατί αν μόνο αντιδρούμε στις σημερινές ε, και χθεσινές πιέσεις, τότε υπονομεύουμε το μέλλον και το, το έργο μας, το μελλοντικό. Άρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε τις δεξιότητες που αναζητούμε, που υπάρχουν. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο οι περικοπές, αλλά να δούμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες, τις προτεραιότητες, τα χρήματα, τους πόρους. Να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί και επ' αυτής της βάσης να τηρήσουμε τα όσα υποσχεθήκαμε. Αλλά χωρίς να ξεχνούμε ότι πρέπει να καταφέρουμε περισσότερα με το δεδομένο προσωπικό περισσότερα και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει σειρά η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση, κυρία Γεωργίευα, ήταν πολύ ωραία και ήταν και γέφυρα, γιατί αυτά θέλαμε εμεί να σας ρωτήσουμε θέματα ανθρωπίνων πόρων ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ο κύριος Ράντεφ, πρώτος από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία ε, Γεωργίευα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έχω την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα και ως Βούλγαρος αλλά και ως Ευρωβουλευτής. Πραγματικά είμαι περήφανος από την ε, δική σας ε, παρουσίαση και σας ευχαριστώ. Ερωτώ λοιπόν, ο κανισμός υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει ότι ε, θα πρέπει να είναι ευρύτερη όσο γίνεται η γεωγραφική βάση για την πρόσληψη ευρωϊπαλλήλων. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες ε, εθνικότητες υπερεκπροσωπούνται. Ενώ το σχετικό ειδικό βάρος άλλων δεν αντανακλάται και υποεκπροσωπούνται. Στις γραπτές σας απαντήσεις έχετε προτάσεις για να μειωθεί αυτή η γεωγραφική ανισορροπία, ας πούμε, ε, ειδικού διαγωνισμούς για τις χώρες που υποεκπροσωπούνται. Τι μέτρα θα λάβετε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Είναι για μένα μεγάλη πρόκληση αυτό το θέμα στο χαρτοφυλάκιο. Χαίρομαι όμως που την αναλαμβάνω, αν την αναλάβω, γιατί πιστεύω ότι το προσωπικό μας είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογο και είμαστε περήφανοι για τους υπαλλήλους μας. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για να αντανακλάτε το σχετικό ειδικό βάρος του πληθυσμού και της επιρροής των κρατών μέλων. Ε, εδώ υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και μεγάλο, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι υπάρχουν κάποιες εθνικότητες τις οποίες ε, δεν ενδιαφέρουν ή δεν ελκύουν ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δεν υποβάλλουν αίτηση ε, για, στους διαγωνισμούς. Και όπως ξέρετε και όπως λέμε, όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πρέπει να πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Άρα εμείς θα πρέπει να πάμε και να οργανώσουμε διαγωνισμούς ε, στις χώρες που υποεκπροσωπούνται και στις ελόγω εθνικότητες. Βεβαίως, δεν είναι αυτό το βασικό μας πρόβλημα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι Το πρόβλημα στην ανισορροπία το έχουμε ε, στα μεσαία στελέχη. Ε, τα ανώτατα και τα κατώτατα έχουν καλή εκπροσώπηση. Οι νέοι λοιπόν είναι καινούργοι πραγματικά νέοι, ε, έχουν πάρα πολύ καλά προσόντα και πολύ ενθουσιασμό, αλλά αρχίζουν από τους χαμηλούς βαθμούς. Ξέρετε επίσης ότι έχουμε παλιά κρατημέλη, νέα κρατημέλη. Ε, και καμιά φορά η εφαρμογή των παλιών κανόνων ε, οδηγεί σε αυτή την υποεκπροσώπηση. Δεν θα το χαρακτηρίζει αρνητική μεταχείριση αυτό, η διάκριση. Ωστόσο, ο νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης θα καταστήσει δυνατό ε, να προάγονται όσοι το αξίζουν πιο γρήγορα. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ. Τώρα εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Γιούρη, αλλά της Επιτροπής Προϋπολογισμών, αλλά η ε, ομάδα μου θεώρησε καλό να με προτείνει να λάβω εδώ το λόγο. Κυρία Επίτροπε, είμαι πεπισμένος ότι θα κάνετε πολύ καλή δουλειά ως αρμόδια επίτροπος και θέλω να σας πω ποια είναι τα τρία σημαντικά για μένα που δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις σας. Ρωτήσαμε δύο φορές πού θα βρείτε τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που έταξε ο Γιούνκερ ως επενδυτικό πρόγραμμα και σε τέσσερις εβδομάδες ε, πρέπει να τα προτείνετε. Μιλήσατε για μόχλευση, πολύ ωραία. Πώς εκτιμάτε τις ε, πιθανότητες αυτό το πρόγραμμα να βρει φρέσκο χρήμα και να κινητοποιήσει για τους ιδίους πόρους στη συνέχεια, είπατε ότι θέλετε να δείτε ποιε δυνατότητε εμεί θέλουμε να μας πείτε προς τα πού πάει η συζήτηση. Και για την κρίση των πληρωμών τέλος μας λέτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που έχουμε, αλλά εμεί θα θέλαμε να σας ακούσουμε να λέτε τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πληρώσει ε, τους λογαριασμούς. Σας παρακαλώ κάντε με ευτυχή, απαντήστε μου συγκεκριμένα. Uh, thank you. Σας ευχαριστώ. Για να προσπαθήσω να σας κάλυψω. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, όχι, δεν θα σας ε, χαροποιήσω γιατί όσον αφορά αυτά τα 300 δις θα ήταν ανεύθυνο να σας πω τι θα πρέπει να γίνει πριν γίνει η σχετική συζήτηση ε, στο νέο σώμα των Επιτρόπων, γιατί είναι κι άλλοι συναρμόδιοι, οι ε, άλλοι έχουν ακόμη περισσότερε αρμοδιότητε γιατί πρόκειται για συλλογική μέθοδο εργασία. Οπότε δεν μπορώ να πω περισσότερα. Πάντω υπάρχει ρόλο μπορεί να παίξει ο κοινωνικό προπολογισμό σε αυτό τη θέση μέτρων τώρα. Όσον αφορά την μόχλευση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων με τρόπο πιο στρατηγικό, πιο εστιασμένο κλπ. Δηλαδή να κάτσουμε να δούμε αυτά τα, τα λεγόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα και να δούμε από την άλλη μεριά τις τεθήσεις προτεραιότητες. Δηλαδή, φτιάχνουμε τις θέσεις εργασίας και τις φτιάχνουμε εκεί που θέλουμε, στο τομείς που θέλουμε. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ανταγωνιστικότητα. Οπότε, άπαξ και εξετάζουμε τα μέσα πολιτικής, αυτά τα εργαλεία ε, από, αυτή την οπτική γωνία, τότε είναι το σωστό. Ε, δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι θα πρέπει να γίνει. Οπότε κατόπιν θα πούμε, με αυτά τα εννέα δις, τι κάνουμε, σε ποιο τομέα, πώς θα φέρουμε την αλλαγή, πώς θα αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων για την απασχόληση. Εξετάζοντα επομένω αυτό το οποίο είναι εξελίξη, όχι το παρελθόν. Τι να σα πω, δεν, δεν, δεν μπορώ να σα χαροποιήσω περισσότερο με αυτά που λέω. Τι να σα πω σε δύο λεπτά. Εγώ πάντω καταλήγω στο ότι δύο λεπτά είναι πολύ λίγα για να καλύψω και χαροποιήσω οποιονδήποτε. Αλλά θα με έχετε πέντε χρόνια ολόκληρα. Thank you, Mr. Duda. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντούντα από το ΣΥΑΡ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Έχω κι εγώ μια παρόμοια ερώτηση. Όπως και εκείνη που έκανε ο βούλγαρος συνάδελφος πριν. Δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνετε έτσι ποια χώρα νοιάζει πολύ αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξέρει πώς θα προσελκύσει ανθρώπους με όσο γίνεται περισσότερα προσόντα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους συμπεριλάβει στο προσωπικό της. Σας ρωτάω λοιπόν, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπάρχει μια ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών χωρών μελών. Πώς θα βελτιώσετε αυτές τις στατιστικές ώστε οι χώρες οι οποίες υποεκπροσωπούνται με προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψουν την διαφορά και συγχρόνως να έχουμε τους καλύτερους υπαλλήλους. Απάντηση. Πράγματι, ο κανονισμός προσωπικού προβλέπει βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί χωρίς βέβαια να πλήττεται η αξιοκρατία, γιατί η αξιοκρατία είναι το βασικό, έτσι, για να έχουμε τους καλύτερους υπαλλήλους. Με το νέο κανονισμό πάντως μπορούμε να έχουμε και δράσεις προκειμένου να μειώσουμε τις ανισορροπίες αυτές. Όντως, η χώρα σας είναι μία από εκείνες η οποία θα έλεγα δεν εκπροσωπείται όσο άλλες. Ίσως γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί Πολωνοί που να είναι υποψήφοι. Πώς θα το διορθώσουμε αυτό. Πηγαίνοντας στα πανεπιστήμια στην Πολωνία, φροντίζοντας το, τα επαγγέλματα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο προσιτά στους πολίτες και η νέα ρύθμιση μας το επιτρέπει αυτό και για την Πολωνία αλλά και για άλλες χώρες. Τα επόμενα χρόνια, μάλιστα όσο συνταξιοδοτούνται περισσότεροι υπάλληλοι, θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά. Και είναι κάτι που θα προσέξω όλους ιδιαίτερος. Γιατί είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι σωστό. Όλοι μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν. Ευτυχώς έχουμε μια υπηρεσία προσλήψεων πάρα πολύ καλή, με ωραίες ιδέες, καλές ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Έτσι λοιπόν θα φροντίσουμε να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία. Αλλά με αξιοκρατία πάντα, έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Χαουτάλα τώρα. Εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ξέρετε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει μια βάση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Πρόκειται για το άρθρο 298 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του άρθρου αυτού είναι η βελτίωση της δίκησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει νομοθεσία η οποία να δεσμεύει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς απέναντι στους πολίτες. Είναι σημαντικό αυτό γιατί όλο όσο περισσότερες εξουσίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο πιο σημαντικό είναι οι πολίτες της να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Δίκηση. Σας ρωτάω λοιπόν, το θέμα αυτό θα το προωθήσετε με τον κύριο Τίμερμαντς. Και παρεπιπτόντως, μιλάμε πολύ για σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να το λύσουμε καλύτερα αν είχαμε καινούργια νομοθεσία. Γιατί βλέπετε τώρα τελικά δεν ξέρουμε καλά καλά τι είναι αυτό που δημιουργεί τη σύγκρουση συμφερόντων. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στις γραπτές μου απαντήσεις το έχω συμπεριλάβει και με τον κύριο Τίμερμανς εφόσον και αυτός επιβεβαιωθεί θα το συζητήσουμε, γιατί πιστεύουμε και οι δύο ότι είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει μια απάντηση. Το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά να τοποθετηθούμε και να αξιολογήσουμε τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 298. Θα έλεγα λοιπόν ότι περιμένω πως και ο κύριος θα το πει. Μόλις αναλάβουμε τα καθήκοντά μας θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε στο Κοινοβούλιο με μια πολύ σοβαρή απάντηση. Ετοιμάζοντας πάντως την απάντησή μας πρέπει πρώτα να δούμε λίγο τι ρυθμίσεις ήδη υπάρχουν, πού υπάρχουν κενά και πώς θα καλυφθούν καλύτερα τα κενά, με ποιο τρόπο γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας χώρος που έχει εξελιχθεί διαφορετικά στο χρόνο. Από την άλλη βέβαια, αυτό που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι ότι πρόκειται για μια νομοθεσία η οποία επηρεάζει μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή τελικά έχει και επιπτώσεις και στις χώρες μέλη. Και αν ναι, τι επιπτώσεις έχει. Και αν ναι, πώς θα αντιδράσουν οι χώρες μέλη. Και για να τελειώσω με αυτό, εγώ πιστεύω πως σήμερα πρέπει να δούμε πόσο θα κοστίσει κάθε λύση, πώς θα ωφεληθούμε και πώς θα έχουμε τη συμμετοχή όλων. Να μην υπάρχουν ε, αποκλεισμοί και να μην φτιάξουμε μια νέα, ένα νέο πεδίο μάχης. Ευχαριστούμε. Τέλος, η κυρία Κομοντίνη από το ΕΛΚ. Κυρία Υποψηφή Επιτροπή, το καταστατικό στο άρθρο 27 ορίζει ότι για να διευκολυνθούν οι προσλήψεις με όσο γίνεται ευρύτερη γεωργική βάση, τα θεσμικά όργανα θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν την ε, γλωσσία όσον αφορά την εκπαίδευση των ε, παιδιών των υπαλληλικών Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στα ευρωπαϊκά σχολεία. Έχουμε σοβαρά προβλήματα να βρούμε ε, αποσπασμένους καθηγητές από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, οικονομικές περικοπές. Εσείς τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα που αφορά και τον χώρο και του διδάσκον προσωπικό και την πρικοδότηση του σχολείου. Τι θα κάνω. Κοιτάξτε, τα οικονομικά προβλήματα, ναι, τα γνωρίζω, είναι σαφή. Έχουμε εδώ μια κατάσταση κατά την οποία πάρα πολύ ωφελούνται από τα ευρωπαϊκά σχολεία όμως μια που είναι ο κοινωνικός προϋπολογισμός που καλεί τα ευρωπαϊκά σχολεία ε, τι να κάνουμε ε, θα πρέπει να πάει κανεί ε, στην Φραγκφούρτη, στην Κεντρική Τράπεζα ε, και να το υποστηρίξει αυτό το, το θέμα το ότι όλοι οφείλονται τα ευρωπαϊκά σχολεία εκεί. Έχουμε στρατηγική, ξέρουμε το πρόβλημα, έχουμε δεσμευθεί, γίνονται ενέργειες. Και εγώ καθώς μια φορά θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσον αφορά τουλάχιστον τα οικονομικά του σχολείου. Και το ίδιο ισχύει και για τις Βρυξέλλες. Μας έχουν έχουμε μια προσφορά τέλο πάντων, πολύ καλή, Όμω είναι 50 χιλιόμετρα μακριά. Δεν θα ωφελήσει και τόσο πολύ όσον αφορά το να λύσουν το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στα ευρωπαϊκά σχολεία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλουμε φυσικά να έχουμε ε, ποικιλία, πολυμορφία, τέλο πάντων, για το προσωπικό αλλά και για την εκπαίδευση, για τις οικογένειες των υπαλλήλων, γιατί ακριβώς είναι κομμάτι του πόσο ελκυστικό να εργάζεται κανείς εδώ. Και συνήθως δεν είναι μόνο τα χρήματα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που κάνουν ελκυστική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολλές φορές ε, Κάνει είναι πιο χαρούμενος στην πατρίδα του, ο ιδιωτικός τομέας δίνει περισσότερα χρήματα, αλλά θέλουμε τώρα να δούμε ότι αυτό το πακέτο το ελκυστικό, πώς ε, φυσικά θα έχει μέσα ως ελκυστική και την εκπαίδευση για να μπορούμε να ελκύσουμε τους νέους που έχουν νέες οικογένειες με παιδιά κλπ. Θα επανέλθω και θα σας πω σε εσά άμεσα, κατευθείαν, όταν μάθω. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίευα. Λέω ο πρόεδρος ε, και εδώ τελειώσαμε τις ερωτήσεις ανεπίτροπη και ξανά έχει τη σκητάλη τώρα ο